Buenos días. Καλημέρα σας. Να ξεκινήσουμε σιγά σιγά την, την συνεδρίασή μας. Σας καλωσορίζω όλες και όλους. Έχετε στους φακέλους αυτό το σχέδιο μέσα της διάταξης. Αν δεν υπάρχει κάποια παρατήρηση για ενδεχόμενη αλλαγή, να σας πω ότι υπάρχει μια αλλαγή. Δεν θα μπορέσουμε να ψηφίσουμε για την δεύτερη, στην προκειμένη περίπτωση, αντιπρόεδρο, διότι η διάσκεψη των πρόεδρων μέχρι στιγμής δεν έχει επιλύσει το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε και το οποίο γνωρίζετε. Στην ε, Επιτροπή μας υπάρχουν μέλη τα οποία δεν είναι τακτικά μέλη της Επιτροπής Εξωτερικών υποθέσεων. Άρα, ουσιαστικά δεν θα έπρεπε να είναι μέλη του Προεδρείου εδώ, στην Υποεπιτροπή μας. Είναι θέμα κανονισμού. Είναι, θα έλεγα, γραφειοκρατικό το ζήτημα. Η κυρία Παγάθα Ορτουντά που την πρώτη ομάδα της για τη θέση της δεύτερης αντιπροέδρου συμμετέχει στις συνεδριάσεις ε, χωρίς πρόβλημα και όταν η διάσκεψη των προέδρων ε, λύσει το διέξοδο θα ολοκληρωθεί το Προεδρείο μας που ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί ακριβώς γιατί δεν εκπροσωπεί τη ομάδα της. Δεν είναι στα δικά μας χέρια όμως, άρα ε, δεν μπορούμε αυτό το σημείο της μερίσιας διάταξης ε, και θα το, να το φέρουμε σε πέρας. Αν δεν έχετε άλλη παρατήρηση, εγκρίνεται η μερίσια διάταξη. Σύντομες ανακοινώσεις τώρα της Προέδρου. Την προηγούμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο εγκρίναμε αρκετά ψηφίσματα για τα κατεπήγοντα, τα γνωρίζετε, είναι και στο πλαίσιο των εργασιών της υποεπιτροπής μας. Και θέματα που θα μας απασχολήσουν και μας απασχολούν ήδη τους επόμενους μήνες, κατάσταση σε Ιράκ και Συρία και η επίθεση του Ισλαμικού κράτους, η δίωξη των μειονοτήτων επίσης, ε, η διωγμή των μειονοτήτων, η κατάσταση στη Λιβύα, την Ουκρανία. Και βέβαια η ανάγκη να υπάρξει μια πιο αποφασιστική απάντηση τη ευρωπαϊκή Ένωση στην επιδημία του Ιέμπολα στη Δυτική Αφρική. Το Προεδρείο, το διευρυμένο Προεδρείο της Επιτροπή μα, είχε την ευκαιρία να συναντηθεί στο πλαίσιο ενός γεύματος εργασίας, αλλά δυστυχώς για ε, λόγους υγείας δεν μπόρεσα να παραστώ. Υπήρχαν πάντως ε, εκεί ε, μεταξύ άλλων ο κ. Λαμπρινίδης, ο εκπρόσωπος Ευρωνώσης για τα θέματα δικαιώματα και άλλοι ε, καλεσμένοι. Είχαμε ενδιαφέρουσες ανταλλαγές απόψεων και στις 13 Οκτωβρίου επιβεβαίωσε ο κ. Λαμπρινίδης ότι θα είναι στη συνεδρίασή μας για ανταλλαγή απόψεων και για να του θέσουμε τα ζητήματα που μας ενδιαφέρουν. Όπως γνωρίζετε, στις τελευταίες συναντήσεις και συνεδριάσεις μας όλοι και όλοι συμφωνήσαμε ότι αυτό που αποκαλούμε business and human rights, επιχειρήσεις και ανθρώπινα δικαιώματα, σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως σε τρίτες χώρες, από τις επιχειρήσεις, από την επιχειρηματική δραστηριότητα, θα είναι ένα βασικό αντικείμενο εργασίας, έρευνας από την Επιτροπή μας και θα διατυπώνουμε σχετικές προτάσεις εξού και έχουμε προβλέψει και σήμερα το πρωί μια κρόαση ακριβώς για το θέμα αυτό. Σεβασμό ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δικαιωμάτων των εργαζομένων εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις επιχειρήσεις, τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Εμένα θα με ενδιαφέρει να δούμε την ευθύνη των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων σε ό,τι αφορά το, τα δικαιώματα των εργαζομένων και τα ανθρώπινα δικαιώματα σε τρίτες χώρες. Νομίζω ότι είναι ένα ζήτημα που δεν το έχει ακόμη ε, εξετάσει επαρκώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στην προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο, βέβαια, εκπονήθηκαν ε, δύο-τρεις εκθέσεις, μία από τον κύριο Χάουιτ, αλλά νομίζω ότι πολύ περισσότερα πρέπει να γίνουν με βάση ε, την αρχή που με διέπει, ότι δηλαδή ε, καλό είναι να δίνουμε το παράδειγμα και όχι και να κηρύσουμε στους άλλους τι πρέπει να κάνουν. Και νομίζω ότι πολλά πρέπει να κάνουμε για να δώσουμε το καλό παράδειγμα και μετά να δίνουμε μαθήματα σε άλλους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε λοιπόν μαζί μας ανθρώπους ε, ειδικούς που εδώ και χρόνια επιτόπου ερευνούν, ε, εξετάζουν το θέμα αυτό. Ήρθε ο πρώτος ομιλητής. Α, ήρθε γιατί ερχόταν από το αεροδρόμιο. Ζιλμπέρ Φουσό Ούγκο. Αναπληρωτής Διευθυντής ε, για τις επιχειρήσεις της Παγκόσμιας Οργάνωσης εργασίας και έπειτα θα δώσω το λόγο σε κάποιους άλλους ειδικού που έχουν έλθει. Θα σας του συστήνω τον καθένα ξεχωριστά όταν έρχεται η ώρα να πάρει το λόγο. Ο Παγκόσμιο Οργάνωση Εργασία ξέρουμε ότι κάνει πάρα πολλή δουλειά, έχει διατυπώσει πάρα πολλέ πολιτικέ, πάρα πολλέ προτάσει για το θέμα αυτό, περισσότερε από οποιονδήποτε άλλο οργανισμό. Και θα δώσω στο τον στον κύριο Φώσου. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα ήθελα καταρχάς να ζητήσω συγγνώμη που έφτασα με μικρή καθυστέρηση. Να σε ευχαριστήσω που καλέσατε το Διεθνή Οργανισμό Εργασίας σε αυτή τη συζήτηση όσον αφορά τις επιχειρήσεις και τα δικαιώματα των εργαζομένων θα ήθελα επίσης να συγχαρώ τα μέλη για την επανεκλογή τους στο Κοινοβούλιο ε, διότι είναι η πρώτη φορά που είχα την ευκαιρία να βρεθώ μπρος σε αυτόν τον χώρο τον επιφανή Εν πρώτης θα ήθελα να αναφέρω βασικά δικαιώματα για τα δικαιώματα των εργαζομένων σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία μετά θα αναφερθώ στα διάφορα εργαλεία τα μέσα που υιοθετήθηκαν το Διεθνές Γραφείο Εργασίας για να αντιμετωπιστούν διάφορα προβλήματα και στο τέλος θα κάνω κάποιες ε, προτάσεις αν μου επιτρέπετε όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα μπορούσαν να συμβάλλουν στο σεβασμό των δικαιωμάτων των εργαζομένων στις αναπτυσσόμενες ε, χώρες. Κυρίες και κύριοι, η ανάγκη για παγκοσμιοποίηση ισότιμη και δίκαιη επιβάλλεται κάθε μέρα και περισσότερο. Η Παγκόσμια Επιτροπή για την Κοινωνική Διάσταση της Παγκοσμιοποίησης που δημιούργησε ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας το 2003 αναφέρει στη σχετική έκθεση ότι οι πολυεθνικές επιχειρήσεις είναι σημαντικότατη φορής αλλαγής στη διαδικασία της παγκοσμιοποίησης αυτές οι επιχειρήσεις τονώνουν την οικονομική ανάπτυξη στις χώρες υποδοχής και παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στη διασυνοριακή μεταφορά κεφαλαίων τεχνογνωσίας, πόρων, τεχνολογίας. Το ότι πρέπει να φροντίσουμε για το σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των αρχών στον χώρο εργασίας είναι κάτι που προσφέρει αδιαμφισβήτητα πλεονεκτήματα και αυτό θα πρέπει να το αναγνωρίσουμε για την ανάπτυξη του δυναμικού του ανθρώπινου και όσον αφορά την οικονομική ανάπτυξη και μπορεί έτσι να συμβάλλει στην οικονομική ανάκαμψη σε παγκόσμιο επίπεδο και στην κοινωνική δικαιοσύνη για μια βιώσιμη ειρήνη η σχετική διακήρυξη που αφορά τις αρχές για τα θεμελιώδη δικαιώματα του 1988 για το χώρο εργασία και για την κοινωνική δικαιοσύνη για μια δίκαιη παγκοσμιοποίηση του 2008 αμοιβαία ενισχύονται και θέλουν να δώσουν μια κοινωνική διάσταση στην παγκοσμιοποίηση και στην πρόθεση της οικονομίας και να οδηγήσουν όλες αυτές οι προσπάσεις σεβασμό των δικαιωμάτων εργαζομένων. Δυστυχώς, οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων πολλαπλασιάζονται. Το βλέπουμε ότι έχει αυξηθεί ο αριθμός των περιπτώσεων που κάθε χρόνο εξετάζονται από την Επιτροπή Συνδικαλιστικών Ελευθεριών ε, του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας. Πέρσι, πέρσι αυτή η Επιτροπή εξέτασε 100 περιπτώσεις υπάρχουν ε, σήμερα στον κόσμο και πρέπει να το υπενθυμίσουμε 168 εκατομμύρια παιδιά που εργάζονται και 22 εκατομμύρια θύματα καταναγκαστικής εργασίας. Τα δικαιώματα των μεταναστών εργαζομένων δεν γίνονται σεβαστά. Η ισότητα ανδρών και γυναικών πόρο απέχει από το να είναι εξασφαλισμένη. Πέρσι η, κα κατάρρευση στη Ράνα Πλάζα, του Ράνα Πλάζα στη Μπαγκλαντές κόστιστε στη ζωή πάνω από, σε πάνω από 1.100 άτομα, κυρίως γυναίκες. Έπληξε τα πνεύματα αυτό το ατύχημα πέρα από τα σύνορα του Μπαγκλαντές και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το ίδιο έκανε διάφορα ψηφίσματα πάνω στο θέμα. Ξέρουμε και το τελευταίο ψήφισμα που πέρασε. Λοιπόν, η οικονομία χαρακτηρίζεται από ανταγωνισμό σε παγκόσμιο επίπεδο και δημιουργούνται μεγάλες αλυσίδες, επικρατούν οι μεγάλοι οικονομικοί φορείς. Και όπως γνωρίζουμε όλοι, πολλά αγαθά και προϊόντα που καταναλώνουμε σήμερα πολύ συχνά κατασκευάζονται σε διάφορα μέρη του κόσμου και είναι αλήθεια ότι όλη η λυσίδα εφοδιασμού παρεμβαίνει σε διεθνές επίπεδο, υπερεθνικό επίπεδο και αυτή η προσέγγιση δημιούργησε θέσει εργασία που χρειάζονται κυρίω στι λιγότερο ανεπτυγμένε χώρε. Ταυτόχρονα όμω, αυτή η αλυσίδα εφοδιασμού δημιουργεί ερωτηματικά όσον αφορά την ποιότητα των θέσεων απασχόληση που δημιουργούνται και όσον αφορά τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Πράγματι, πολλέ πρόσφατε τραγωδίε συνδέονται με την εργασία και θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί αν οι εθνικέ προδιαγραφέ και διεθνεί παρόμοιες ε, είχαν τεθεί σε ισχύ, ίσια. Αλλά είναι πολύ περίπλοκο το σύστημα εφοδιασμού. Οι συνθήκες εργασίας και επαγγελματικέ ε, σχέσεις βέβαια ρυθμίζονται νομικά από εθνική νομοθεσία. Δυστυχώς ε, σε πολλές χώρες με χαμηλό εισόδημα και θα έλεγα ακόμα σε κάποιες χώρες μέσου εισοδήματος που διαθέτουν όμως θεσμικό δυναμικό, αρκετά δύναμο, ή μειωμένο πλαίσιο θεσμικό, σε αυτές τις χώρες η εφαρμογή του νόμου, πώς να το πω στα αγγλικά, η επιβολή του νόμου, της εθνικής νομοθεσίας, ε, αποτελεί μεγάλη πρόκληση και δυσκολία και κάποιες αλυσίδες εφοδιασμού όπως τα έτοιμα ενδύματα ε, συνεχώς ε, πολλαπλασιάζουν τι υπεργολαβίες. Υπάρχει τόσο μεγάλο επίπεδο υπεργολαβίες που φτάνει στο να απασχολεί πολύ μικρές επιχειρήσεις. Και είναι πολύ δύσκολο σε αυτές τις πολύ μικρές επιχειρήσεις να μπορεί να επιβάλλει κανείς τα δικαιώματα των εργαζομένων. Δεν μπορούμε όμως να γνωρούμε ε, τις θέσεις που προσφέρονται, κυρίως από τους βασικούς φορείς, ε, διότι πρέπει να υπάρχει αστερός έλεγχος των προϊόντων, κυρίως των προϊόντων που πολλούνται με το, η μεγάλη παραγωγή, πρέπει να ελέγχουν καλύτερα τα προϊόντα συνθήκες στις οποίες ε, εργάζονται. Πρέπει να υπάρξουν νέες συμφωνίες με εργαζομένους κυβερνήσεις και εργοδότες και στις χώρες που καταναλώνουν και στις χώρες που παράγουν. Χρειάζεται αυτή η βάση. Λοιπόν, το Διεθνέ Γραφείο Εργασίας, μαζί με διεθνείς ε, με φορείς που σχετίζονται με την Παγκόσμια Τράπεζα, ξεκίνησε ένα πρόγραμμα που γνωρίζετε αρκετά καλά, ε, που είναι ένα πρόγραμμα που αφορά την επιβολή καλύτερων συνθήκων εργασία, λέγεται Better Work. Ε, στόχο είναι η βελτίωση τη ανταγωνιστικότητα των θέσεων απασχόληση στο παγκόσμιο εμπόριο, χάρη σε προγράμματα εθνικής εμβέλειας στον τομέα της ένδυσης. Ε, νομίζω ότι συμπράξεις που δημιουργούνται τέτοιου τύπου ε, δημιουργούν κάποιες ελπίδες για τις γυναίκες και τους άντρες που εργάζονται και που χρειάζονται, έχουν μεγάλη ανάγκη μεγαλύτερης προστασίας. Το Εθνές Γραφείο Εργασίας είχε θετήσει και τη διακήρυξη την τριμερή των αρχών ε, όσον αφορά την κοινωνική πολιτική πρέπει να ακολουθείτε και πιστεύουμε ότι είναι πάρα πολύ επίκαιρο αυτό το πλαίσιο. Είναι ένα μέσο αυτή η διακήρυξη και θεωρεί ότι οι επαγγελματικέ σχέσει, η συνδικαλιστική ελευθερία και οι συλλογικέ διαπραγματεύσει, όλα αυτά αποτελούν μέσα για την επίτευξη θετικών αποτελεσμάτων. Όταν χρησιμοποιείται πλήρω, προωθούνται άριστα τα δικαιώματα των εργαζομένων σε παγκόσμια κλίμακα. Βασικά, αν η αλληλεγγύη, κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων και η τεχνική βοήθεια είναι, τεχνικά, είναι μάλλον ε, σημαντικά, αλλά χρειάζεται και πλαίσιο θεσμικό, σαφές, δίκαιο, ε, με ένα σύστημα εφαρμογής που θα είναι πατολεσματικό όσον αφορά την επιβολή της νομοθεσίας και θα πρέπει οι εθνικοί θεσμοί να επιτρέπουν στους κοινωνικούς εταίρους να παίξουν πλήρη, ρόλο, ούτως ώστε να σημειωθεί πραγματική πρόοδος ε, που θα είναι και βιώσιμη εντάχει. Κλείνοντας, θέλω να διατυπώσω αξιότιμοι κύριοι βουλευτές κάποιες ε, προτάσεις, συστάσεις. Εμπρότης, φρονών την απαραίτητο να συνεχιστεί το έργο ευαισθητοποίησεως όσον αφορά αυτά τα θέματα και εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα πλαίσια σχέσεων Ευρωπαϊκής Ενώσεως με τον εξωτερικό κόσμο. Είμαι βέβαιος ότι πολλοί από εσά ήδη συμμετέχετε ενεργά στην προσπάθεια και αυτές οι προσπάθειές σας θα έχουν συνέχεια. Είδα θετικό αντίκτυπο ήδη των πιέσεων της εκστατείας ευαισθητοποίησεως ε, που προέρχεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μετά τρίτον, στις σχέσεις σας με άλλες χώρες, στο διάλογό σας που έχετε με αυτές για τα ανθρώπινα δικαιώματα θα μπορούσατε να λάβετε υπόψη την ανάγκη να υπογραμμιστεί η σημασία της συμμόρφωσης των εθνικών νομοθεσιών και των διεθνών προγραφών εργασίας με τη συνδυαστική ελευθερία και την ελευθερία των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Τρίτον, σε πολλές αναπτυσσόμενες χώρες, όπως προανέφερα, το θέμα της εφαρμογής των μέτρων από τη στιγμή που η εθνική νομοθεσία έχει υιοθετηθεί, μέσω έγκρισης διεθνών συμβάσεων, έλεγα η επιβολή όλων αυτών των νόμων αποτελεί πρόκληση. Το υπενθύμησα προηγουμένω αυτό. Δεν εφαρμόζονται σωστά οι νόμοι. Και μπορεί να γίνει αυτό θέμα συνεργασίας στα πλαίσια της αναπτυξιακής βοήθειας. Μπορείτε να το εξετάσετε αυτό, ναι, σε ποιο βαθμό σε αναπτυξιακά προγράμματα που εφαρμόζονται διάφορες χώρες μπορείτε να εντάξετε και ε, την εφαρμογή των νόμων που ήδη έχουν θεσπιστεί. Τέταρτον, κλείνοντας εδώ, θα μπορούσατε να θέσετε και το θέμα της οικονομικής και τεχνικής βοηθείας που είναι απαραίτητες για να εξασφαλιστεί μια αποτελεσματική εφαρμογή των διεθνών προδιαγραφών στα κεφάλαια τα σχετικά με την βιωσιμότητα των συμφωνιών ελευθέρων συναλλαγών που υπογράφει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τρίτες χώρες. Ιδού λίγο πολύ οι θέσεις που ήθελα να σας παρουσιάσω και σταματώ εδώ ευχαριστώντας σας κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Ουγμπό. Αργότερα θα έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε μαζί σας και με τα μέλη της Επιτροπής μας. Και τώρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Στίβεν Μπένετικτ, που και αυτός έφτασε τελευταία στιγμή. Είναι διευθυντής δικαιωμάτων ε, των ανθρώπων και συνδικάτων από την Διεθνή, από την Ένωση των Διεθνών Συνδικάτων. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αν με επιτρέπετε θα μιλήσω αγγλικά. ευχαριστώ καταρχάς που με προσκαλέσατε να δώσω τη μαρτυρία μου ενώπιον της Επιτροπής σας. Θα ήθελα λοιπόν να πω κατευθείαν στην ουσία και να αναφερθώ στις προοπτικές της ε, Διεθνούς Συνδικαλιστικής Ένωσης και τα σχόλια σε σχέση με τα όσα ήδη είπε ο γενικό Διευθυντής τη ε, παγκόσμιου Οργάνωση Εργασία κ. Χούμπο. Ασφαλώς, τα ανθρώπινα δικαιώματα σε πολλές περιοχές του κόσμου ε, παρουσιάζουν οπισθοδρόμηση. Η έρευνα τη Διεθνού Νομοσπονδίας μας, ITUC, για τις, παραβιάσεις των δικαιωμάτων που σας έχω φέρει και σε αυτό το εγχειρίδιο δείχνει ξεκάθαρα ότι τα εργασιακά δικαιώματα πλήττονται τόσο από τις επιλογές των κυβερνήσεων που προσπαθούν να περιστύλουν με την νομοθεσία τα δικαιώματα των εργαζομένων, όσο και από τους εργοδότες οι οποίοι παραβιάζουν τα δικαιώματα ατιμωρητοί. Πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να διαδραματίσει πλήρω το ρόλο που τη ανήκει στην οικονομική και την κοινωνική πολιτική, έτσι ώστε να εξασφαλίσει ένα περιβάλλον μέσα στο οποίο θα μπορούν άφοβα να ασκούν και να διεκδικούν τα δικαιώματά του οι εργαζόμενοι. Έμφαση έχει ορθά τεθεί ως προς την αντιμετώπιση του ζητήματος της ε, κλιματικής αλλαγής και εδώ θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ε, επιχειρήσεις οι οποίες εδρεύουν σε αυτήν έχουν ιδιαίτερο ρόλο. Θα πρέπει δηλαδή να βεβαιωθούν ότι όσοι εργάζονται ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για την Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να μπορούν να κερδίσουν τα προστοζήν μέσα σε μια εβδομάδα εργασίας με λογικά ωράρια με λογική διάρκεια. Θα ήθελα πολύ στόμα λοιπόν να αφαιρθώ σε τρεις χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας και ίσως στη διάρκεια της συζήτησης να επεκταθώ και στη Γουατεμάλα προς το παρόν όμως θα περιοριστώ σε αυτές τις τρεις χώρες. Βυρμανία, Μιαρμάρ. Καθώς τώρα έρονται οι εμπορικές κυρώσει που ίσχυαν επί πολλά χρόνια βάρο τη ε, χώρα Έχουμε μια σειρά από επιχειρήσει από τις ΗΠΑ στην Ευρώπη αλλά και από άλλε περιοχέ του κόσμου που εγκαθίσανται στη χώρα αυτή. Είναι ασφαλώ αυτονόητο το γιατί θεωρείται τόσο ελκυστική τώρα η Βυρμανία. Θεωρείται ότι είναι ο κύριο πλέον ή ο, ο ε, ε, χαμηλού κόστους εργατικού δυναμικού του κόσμου, ο προσεχής κόμβος μετά τον Μπαγκλαντές για τις μεγάλες επιχειρήσεις. Η Βυρμανία ασφαλώς και χρειάζεται επενδύσεις. Πλην όμως οι επενδύσεις αυτές θα πρέπει να γίνονται με τρόπο υπεύθυνο, με λογοδοσία και να εξασφαλίζουν μια οικονομική ανάπτυξη με όσο δυνατόν ευρύτερη ε, διανομή των ε, ωφελών. Έτσι λοιπόν χρειάζεται για τη Βυρμανία ένα κράτος στηριζόμενο στο κράτος δικαίου, ενώ τώρα ακόμα παραμένουν πάρα πολλά προβλήματα, ενώ ακόμα ανήκουν στο στρατό ο οποίος διαχειρίζεται το μεγαλύτερο μέρος του πλούτου της χώρας άμεσα ή έμεσα και ενώ πολλές επιχειρήσεις έχουν απλώς καταργήσει τα συνδικαλιστικά σωματεία. Ενώ δε η νομοθεσία ε, για την διευθέτηση εργασιακών διαφορών και για την θέσπιση εργατικών σωματείων υφίσταται, έχει θεσπιστεί, ε, πράγμα για το οποίο βεβαίω εκφράζουμε την ικανοποίησή μας, Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα και κενά και ως προς την άσκησή της, προς την υλοποίησή της και διατάξεις οι οποίε παραβαίνουν το διεθνέ δίκαιο. Επιπλέον, διοικητικό ή ε, δικαιοδοτικό σύστημα το οποίο να εξασφαλίζει την ε, ουσιαστική υλοποίηση της νομοθεσίας αυτής δεν υπάρχει. Και μάλιστα αυτή η απουσία κράτους δικαίου παραμένει σοβαρότατο πρόβλημα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναγνωρίσει, αναγνωρίσει ήδη ότι θα πρέπει οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να τηρούν πολύ αυστηρά πρότυπα υπεύθυνων επενδύσεων όταν αναλαμβάνουν δραστηριότητες και επενδύουν στην Βιρμανία. Τον Ιούνιο του 2013 η Επιτροπή Άστον και το αναφερόμενη στην επανεισαγωγή του γενικευμένου συστήματος προτιμήσεων ε, δήλωναν ότι οι υπεύθυνε επενδύσει και το διμερές εμπόριο είναι στοιχεία απαρέγκλητα για την ανάπτυξη και την ανάκαμψη του εμπορίου. Δήλωση η οποία αντικατοπτρίζει ε, δηλώσεις του Συμβουλίου του Απριλίου του 2012 για υπεύθυνες δραστηριότητες των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στη Βιρμανία Μιανμάρ, οι οποίες θα πρέπει να προάγουν την πρακτική των ύψιστων προτύπων ακεραιότητας και υπεύθυνη επιχειρησιακής δραστηριότητας και ιδιαίτερα αυτό αναφερόταν στις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, τις ε, κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υπεύθυνη επιχειρησιακή στρατηγική 2011-2014. Πλην όμως, Μέχρι τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει δώσει ιδιαίτερη ε, βάση σε αυτές τις δηλώσεις, δεν έχει μετατρέψει σε έργα αυτές τις δηλώσεις. Από την άλλη έχουν αναλυφθεί κάποια μέτρα για την προαγωγή υπεύθυνων επενδύσεων με την έκδοση νέων υποχρεώσεων για λογοδοσία και ενημέρωση ως προς την υπεύθυνη, της υπεύθυνης επενδύσης στη Βιρβανία από τις ΗΠΑ. Οι αμερικανικές δηλαδή επιχειρήσεις κάθε χρόνο και δημόσια θα πρέπει να ανακοινώνουν μεταξύ άλλων τι είδους επιχειρησιακές δραστηριότητες έχουν στην ε, Βιρμανία, τι είδους ε, πληρωμές καταβάλουν σε κρατική κρατικές, ε, σε κρατικούς φορείς και κατά πόσον υπάρχουν ζητήματα νομοθεσίας εργασιακής κατά της διαφθοράς, κατά της, ε, για την καταπολέμηση της ε, ρήπανσης του περιβάλλοντος και ούτε καθεξής. Και επίσης δημοσιεύεται ένας κατάλογος των ατόμων που αποκλείονται από τη δραστηριότητα στις περιπτώσεις αυτές για λόγους κακής συμπεριφοράς. Θέλουμε λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση τουλάχιστον να έχει ισοδύναμες ε, με αυτές των ΗΠΑ διατάξεων αφορά την επιχειρησιακή δραστηριότητα στη Βυρμανία ώστε να έχουν οι, Ευρωπαϊκέ οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις εξίσου υπεύθυνη συμπεριφορά και θέλουμε μέσα τα οποία θα είναι αντίστοιχα, θα είναι όπως ε, των Ηνωμένων Εθνών, δηλαδή κατευθύριες αρχές ε, των Ηνωμένων Εθνών ή του ΟΣΑ ή αρχές ή οι δηλώσεις του, ε, της Διεθνής για την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα. Επίσης θέλουμε να καταγράφεται κάθε είδους συνέπεια για τα ανθρώπινα δικαιώματα από την ανάπτυξη μιας επιχειρηματικής δραστηριότητας, μιας επενδύσεως, καθώς και τα μέσα διευθέτησης διαφορών, πράγμα το οποίο ουσιαστικά θα εξασφαλίζει ότι νέε επενδύσει, νέε συναλλαγέ, δεν θα επιδεινώνουν τα προβλήματα της χώρας και σε κάθε στάδιο θα πρέπει επιχειρήσει, οι οποίες επενδύουν ή δραστηριοποιούνται στη Βυρμανία θα πρέπει να αναγνωρίσουν λοιπόν ότι ε, οφείλουν να συνεργάζονται ανοιχτά και με τρόπο ειλικρινή ε, και με τα συνδικαλιστικά σωματεία. Ε, μία ακρόαση από το Κοινοβούλιο για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στη Βυρμανία πιστεύω θα μπορούσε να δώσει πολύ καλά στοιχεία στο Κοινοβούλιο και στη δημοσιότητα για το ποιες είναι οι επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται εκεί και βεβαίως να πιέσει για τα θέματα των ανθρωπινών δικαιωμάτων και τις στήριξή του στη Βυρμανία. Πολύ σύντομα θα αναφερθώ τώρα στην Καμπότζη. Όπως γνωρίζετε η Ευρώπη είναι μια σημαντική ε, ε, ένα σημαντικός χώρος εξαγωγών προς την, ε, της Καμπότζης, για την Καμπότζη. Έχουμε 1,8 δισεκατομμύρια δολάρια εξαγωγές από την Καμπότζη προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για τους πρώτους 11 μήνες του 2013. Αύξηση σημαντική στην αντίστοιχη περίοδο του σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012 και τάσεις οι οποίες δεν φαίνεται να αντιστρέφονται για το 2014. Εμπόριο λοιπόν ειδών ενδύσεων, ενδύσεως, το οποίο έχει να κάνει και με το ε, σύστημα τα πάντα πλην όπλων για τις ε, πλέον φτωχές χώρες, το οποίο έχει προσπογράψει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Για τις εμπορικές δεπροτιμήσεις έχει εισαγάγει σημαντικές διατάξεις η Ευρωπαϊκή Ένωση που απαιτεί από τον φιλοφελούμενο να τηρεί αυστηρέ προδιαγραφές και πρότυπα εμπορικά. Ωστόσο, η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας έχει επανειλημμένως και επί σειρά ετών καταδικάσει και επικρίνει την Καμπότζη, διότι δεν προάγει την ελευθερία του, συνε... του η κυβέρνηση της ε, Καμπότζης μάλιστα πριν από ένα διάστημα είχε χρησιμοποιήσει πάρα πολύ σκληρή βία κατά διαδηλωτών όταν ε, οι αντιδράσεις των εργατών ε, προκλήθηκαν από την ανακοίνωση νέου κατώτατου μισθού. Υπήρξαν πολλές διαδηλώσεις και αυστηρή καταστολή παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις από μια σειρά ομάδων, φορέων, μη κυβερνητικών οργανώσεων, συνδικαλιστικών σωματείων. 31 εργαζόμενοι παρέμειναν φυλακισμένοι επί εξάμηνο χωρίς τη δυνατότητα υπό όρους αποφυλάκησης, παρότι ορισμένοι από αυτούς χρειάζονταν κατεπηγόντως ιατρική περίθαλψη. Δυστυχώς η κυβέρνηση συνεχίζει, συνεχίζει μια πορεία για ένα ε, νόμο εργατικό που αποτελεί σημαντική όπιστο δρόμη σε σχέση με την υφιστάμενη εργατική νομοθεσία και ο οποίος εφόσον υιοθετηθεί θα περιστείλει ακόμη περισσότερα τα δικαιώματα των εργαζομένων και των ανεξάρτητων συνδικαλιστικών σωματείων. Εάν λοιπόν θέλει ε, Εάν λοιπόν θέλουν οι εργασιακέ διατάξει του ε, συστήματο γενικευμένων προτιμήσεων να ε, φέρνουν ουσιαστικά αποτελέσματα πρέπει και να εφαρμόζονται ουσιαστικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να αντιμετωπίζονται με σοβαρότητα. Η Διεθνή Οργάνωση Συνδικαλιστικών Σωματείων όπω και η Ευρωπαϊκή, ITUC και ETUC, καλούν την Ευρωπαϊκή Ένωση να διαπραγματευτεί ένα σύμφωνο βιωσιμότητα με την Καμπότζη όπω έχει πράξει και με τον Μπαγκλαντές τα εργασιακά δικαιώματα, εφόσον τηρηθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα έχουν σαν αποτέλεσμα ότι ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση αναλαμβάνει τον ηγετικό ρόλο που χρειάζεται σήμερα να αναλάβει και μπορεί έτσι να βοηθήσει στη διοχέτευση πόρων και δυνατοτήτων σε ένα πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων που θα μεταλλάξει τη χώρα και θα είναι ασφαλώς πολύ καλύτερο από ότι μια εμβαλωματική προσέγγιση. Ελπίζουμε λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορεί τώρα να αναλάβει δράση, όπως έπραξε και στο Μπαγκλαντές, ε, εφαρμόζοντας τους δικούς της νόμους, τις δικές της πολιτικές και να μην περιμένει να ε, συμβεί κάποια κάποιο άλλο τραγικό ατύχημα. Ε, όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, η πιο σημαντική πρωτοβουλία για, την συνέχιση, για τη συνέχεια που δόθηκε στην κατάρρευση του κτηρίου του Μπαγκλαντές στο Ράνα Πλάζα ήταν η εξέταση των συνθήκων εργασίας με συμμετοχή πάνω από 2.000 φορέων και εργατικών σωματείων, Ηνωμένε Πολιτείε Ευρωπαϊκή Ένωση, Διεθνής Οργάνωση Εργασίας, μαζί με μια πρόταση για ένα σταθεροποιητικό πρόγραμμα εξασφαλίζουν σημαντική πρόοδο αλλά παρά τα μέτρα αυτά είναι πολύ δύσκολο για τον εργαζόμενο να ασκήσει τα βασικά του εργασιακά δικαιώματα στον Μπαγκλαντές. στις ε, δε ζώνες παραγωγής προϊόντων που απευθύνονται στην ε, εξαγωγή, που προορίζονται για εξαγωγές, απαγορεύονται, απαγορεύεται ο συνδικαλισμός ακόμη στο Μπαγκλαντές. Εδώ έχουμε να κάνουμε έναν τρόπο παραγωγής ο οποίος δεν μπορεί να είναι βιώσιμος, απλώς θα οδηγήσει σε περαιτέρω τραγωδίες. Η απουσία λοιπόν πολιτικής ε, βούλησης ή η αποτυχία της διακυβερνητικής συνεργασίας, τα, υψηλά επίπεδα διαφθοράς, η εμπλοκή, η διαπλοκή ε, του τομέα της κλωτοστοϊφαντουργίας μέσα στην κυβέρνηση οδήγησαν στις καταστροφές ε, του 2012, οι καταστροφές 2012-2013 να μην έχουν πολύ σημαντικές, να μην οδηγήσουν πολύ σημαντικές ανατροπές. Εμείς θα θέλαμε με το σύμφωνο αυτό της βιωσιμότητας να καταγραφεί και η απουσία προόδου και να ε, ενημερωθεί η κυβέρνηση του Μπαγκλαντές ότι πρέπει να αναλάβει δράση ταχύτατα και αποφασιστικά εάν θέλει να αποφύγει τι συνέπειε τη αδράνεια τη. Όπω συμβαίνει και με την Καμπότζη, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αναλάβει μέτρα ώστε να βεβαιωθεί ότι η διεθνή κοινότητα συμμορφώνονται προ τι ευθύνε τη και εξασφαλίζει ένα περιβάλλον μέσα στο οποίο τα δικαιώματα των εργαζομένων σε ολόκληρη την αλυσίδα της προσφοράς ε, την χάνουν σεβασμού. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Ρεμπίκα Σμιθ, η οποία είναι Σύμβουλο, Ανώτερη σύμβουλο για θέματα κοινωνικών υποθέσεων του Business Europe. Παρακαλώ. Ναι. Ευχαριστώ πολύ, ε, κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω την Επιτροπή που κάλεσε την Business Europe σήμερα στην πολύ σημαντική αυτή ακρόαση. Για μα το θέμα είναι σημαντικό και από ό,τι κατάλαβα θα οργανώσετε μια σειρά σεμιναρίων για τα ζητήματα αυτά και η Business Europe θα ήθελε να συμμετάσχει σε αυτές τις συζητήσεις. Θα σας ε, κάνω μια γενική παρουσίαση. Δεν είμαι η Δήμων για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε αντίθεση με άλλα μέλη του πάνελ. Πρέπει να σας πω βέβαια ότι συζήτησα με διεθνείς οργανισμούς, ε, υπαλλήλου αυτών των ε, οργανισμών που ασχολούνται με αυτά τα θέματα σε διεθνές επίπεδο κατά την προπαρασκευή της ομιλίας μου και με άλλους που ασχολούνται με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Καταρχάς να πω ότι η μεγάλη, η τεράστια πλειοψηφία των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε αναπτυσσόμενες χώρες ε, φέρουν ωφέλη στην οικονομία και την κοινωνία, θέσεις εργασίας, παροχή αγαθών και υπηρεσιών, τοπικά συμβόλαια για τις τοπικές επιχειρήσεις. Φυσικά και υπάρχουν ε, ελλείψεις σε διάφορες χώρες και αυτό το έχουμε εντοπίσει, ιδίως στον τομέα των συνθήκων εργασίας. Εν γέννη όμως θεωρούμε ότι το άνοιγμα ε, του εμπορίου των επενδύσεων δίνει την ευκαιρία για ανάπτυξη αυτές τις χώρες και αυτό μπορεί να ωφελήσει και τον πληθυσμό. Οι εταιρείε βέβαια έχουν ε, πολλές ευθύνες απέναντι καταναλωτές, εργαζομένους, μετόχους, άλλους επενδυτές, ε, τις κυβερνήσεις, τις τοπικές κοινωνίες και ούτω καθεξής. Η διοίκηση των επιχειρήσεων πρέπει να λαμβάνει καθημερινά αποφάσεις ε, για να έρθει το ύψος ε, των ευθυνών και των περιστάσεων. Και πολλοί γνωρίζουν ότι η επιτυχία των επιχειρήσεων βασίζεται και στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνών στις οποίες δραστηριοποιούνται. Και αυτό ισχύει και στη χώρα και σε διεθνέ επίπεδο. Πρέπει βέβαια να τηρούν οι επιχειρήσει του νόμου των κρατών ε, όπου δραστηριοποιούνται. Έχουν και ηθική ευθύνη όμω όταν επενδύουν σε αναπτυσσόμενες χώρε. Λαμβάνω σοβαρά το θέμα αυτό. Έξω και πολλέ εταιρείε έχουν ηθικά πρότυπα και κανόνε που εφαρμόζουν σε παγκόσμιο επίπεδο και μέσω τη κοινωνική εταιρική ευθύνη και τη σχετική πολιτική πολλέ επιχειρήσει συμπεριλαμβάνουν και ε, πολλέ ε, ε, περιβαλλοντικές ε, μέρημνες και κοινωνικά ζητήματα στις, ε, στη δραστηριότητά τους. Επίσης το θέμα της, του παγκόσμιου εφοδιασμού, της αλυσίδας εφοδιασμού και το πώς δραστηριοποιούνται και επιχειρήσεις είναι ένα θέμα που θα μας απασχολήσει γενικώ. Και αυτό είναι άκρος πολύπλοκο, ιδίω για επιχειρήσεις που δραστηριοποιείται σε χώρες που η νομοθεσία για τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα δεν εφαρμόζεται ή δεν επιβάλλεται ε, και νομίζω ότι θα πρέπει η πολυπλοκότητα αυτή να ληφθεί υπόψη. Οι επιχειρήσεις αυξάνουν ε, τη συνεργασία τους ε, ε, με τη στρατηγική για την κοινωνική εταιρική ευθύνη και πολλές επιχειρήσεις έχουν δεσμευτεί να προσχωρήσουν σε διεθνείς πρωτοβουλίες ε, ή σε θελοντικές πρωτοβουλίες, παραδείγματος χάρη ανάπτυξη κωδικών δεοντολογίας, καλή συμπεριφορά κτλ. Το βασικό σημείο όμως, που, το βασικό μήνυμα που θέλω να περάσω σήμερα είναι ότι εμείς είμαστε πεπισμένοι ότι οι πολυεθνικές μπορούν να δώσουν ένα ε, μέρος της λύσης και της απάντησης στο θέμα του σύμφωνα των ανθρωπινών δικαιωμάτων θα πρέπει να είναι μέρος αυτής της συζήτησης καθότι είναι και πρωταγωνιστική φορή ό,τι αφορά την οικονομική ανάπτυξη, σώμενο κόσμο. Πιστεύουμε ότι μπορούν ε, να, έχουν μια θετική συνεισφορά σε χώρε με αδύναμη διακυβέρνηση, αυξάνοντα κοινωνικά πρότυπα την ευημερία, βελτιώνοντα επίση και την εκπαίδευση. Βέβαια, είναι σαφέ ότι οι επιχειρήσει δεν μπορούν να επιλύσουν από μόνε τα προβλήματα, διότι δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο ενό νομικού περιβάλλοντο ε, που το δημιουργούν τα κράτη. Και τα κράτη είναι αυτά που πρέπει να ε, μεριμνούν για την εφαρμογή και την επιβολή των νόμων από όλου και να έχουν του κατάλληλου αποπτικού και εφαρμοστικού μηχανισμού. Έρχομαι στο πλαίσιο του Τζον Ρόγκη για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εδώ υπάρχει μια σαφή διάκριση μεταξύ Τη ανάγκη ε, για σεβασμό των θερμιλιωδών δικαιωμάτων και της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης. Η ε, οργάνωση ε, εργαζομένων έχει επίσης ε, ε, συνεργαστεί άμεσα με την Ευρωπαϊκή Ένωση για να τηρηθούν οι κατευθυντήριε γραμμέ των ΗΠΑ και τα σχετικά πρότυπα για το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τη επιχειρήση και συνεργάζονται για την υλοποίηση αυτού του πλαισίου και των κατευθυντηρίων γραμμών σε συνεργασία με το Business Europe. Και αυτό δείχνει και τη δέσμευση του Business Europe. Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές τώρα του ΟΗΕ είναι στη φάση τη εφαρμογή τη υλοποίησης και για ένα είναι πολύ σημαντικό οποιαδήποτε δράση αναλαμβάνεται είτε σε εθνικό, ενωσιακό ή διεθνές επίπεδο να μην θέτει σε κίνδυνο την εφαρμογή αυτών των αρχών. Σε αυτό το πλαίσιο λυπούμεθα που κάποιε χώρε έχουν προτείνει την ανάπτυξη ενό νομικού δεσμευτικού πλαισίου για τη ρυθμίση ε, του κόσμου της διασυνοριακής συνεργασίας έχει ε, επιτευχθεί σημαντική πρόοδο τα τελευταία χρόνια για την υλοποίηση των κατευθυντηρίων αυτών οδηγιών. Θα πρέπει να θυμόμαστε βέβαια ότι μόλις τρία χρόνια έχει ξεκινήσει η διαδικασία αυτή και στην αρχή της ποτέ δεν είχαμε φανταστεί ότι μετά από μια τριετία θα είχαν λυθεί όλα τα προβλήματα φυσικά. Έχουμε εξελίξεις, έχουμε την ανάπτυξη διεθνών ε, προγραμμάτων εργασίας, θα γίνει και μια θεώρηση από στον των σχεδίων δράση και από πλευρά επιχειρήσεων καταρτίζονται πολιτικέ, έχουμε συστήματα αναφορά, ε, δημιουργία υποδομών, ικανοτήτων. Είμαστε στη σωστή κατεύθυνση, στο σωστό δρόμο. Φυσικά και μπορούν να γίνουν περισσότερα. Ένα περιβάλλον αξιόπιστο που θα δίνει δυνατότητε για το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι αυτό που θέλουμε να δούμε. Πιστεύουμε επίση ότι θα πρέπει να καταβληθούν περισσότερε προσπάθειε για να στηριχθούν εκείνα τα κράτη που δεν είναι σε θέση να μεταφέρουν στο εθνικό δίκαιο τι διεθνεί συμβάσει ανθρωπίνων δικαιωμάτων, άλλε συμβάσει για δικαιώματα εργαζόμενων κτλ. Να του δοθεί επίση πρέπει και κατάλληλη τεχνική βοήθεια για να αναπτύξουν τι ε, νομικέ και διοικητικέ δομέ. Πολλέ ευρωπαϊκέ χώρε έχουν ε, ήδη εγκρίνει ή είναι στη φάση τη έγκριση εθνικών σχεδίων δράση. Και υπάρχει η ομάδα εργασία του ΟΗΕ ε, για τα εθνικά αυτά σχέδια δράση που μπορεί να βοηθήσει και να ενισχύσει τι προσπάθειε αυτών των χώρων και να εμπνεύσει και άλλε χώρε να πράξουν το ίδιο. Έχουμε και τη Διεθνή Οργάνωση Επιχειρήσεων ε, της Αφρικής που αναφέρει τα πλεονεκτήματα της κατάρτισης σχεδίων εργασίας και παροτρύνει τα κράτη να λαμβάνουν πολύ σοβαρά τις δεσμεύσεις του. Σίγουρα υπάρχουν τεράστιες διαφορές μεταξύ των χωρών. Πρέπει να υπάρχει ευελιξία. Κάθε χώρα να επιλέγει τα πλέον κατάλληλα εργαλεία πολιτικής για να αντιμετωπίσει τη συγκεκριμένη κατάσταση που ισχύει στην εκάστοτε χώρα. Και βέβαια δεν σταματάει η κατάρτιση σχεδίων δράση με την έγκρισή του. Υπάρχουν χρονοδιαγράμματα και για την αξιολόγηση των εθνικών αυτών σχεδίων δράση. Τώρα, να πω λίγα λόγια και με αυτό θα ολοκληρώσω για τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας. Πάνω από 180 συμβάσεις ε, και πάνω από 200 συστάσεις ε, έχουν διατυπωθεί από, τον, ε, από τη Διεθνή Αυτή Οργάνωση Εργασίας. Υπάρχει, είναι ένας τριμερής επίσης οργανισμός αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο του Διεθνούς, της Διεθνής Οργάνωσης για την εκπόνηση προτύπων. Και όσες χώρες προσχωρούν σε αυτές τις συμβάσεις πρέπει να εφαρμόζουν τις συστάσεις και τις διατάξεις, να αναφέρουν για την εφαρμογή. Υπάρχουν και ε, μηχανισμοί ε, καταγγελιών, προσφυγών, σε περίπτωση που μια χώρα παραβιάσει τις συμβάσεις που έχει επικυρώσει. Πρέπει να θυμόμαστε ότι οι συμβάσεις ε, της ΔΟΕ εφαρμόζονται σε χώρες. Ίσως να μην είναι απάντηση σε όλα τα προβλήματα που υπάρχουν στον εργασιακό κόσμο και χώρο. Θα πρέπει να μπορούν όμως να επηρεάζουν εκεί που έχουν ένα μεγάλο αντίκτυπο και θα πρέπει να υπάρχει και συνένεση σε επίπεδο ΔΟΕ για να μπορούν να προωθηθούν ορισμένα μέτρα. Επίσης θα πρέπει να υπάρχουν ε, κατώτατοι ελάχιστοι κανόνες που να μπορούν να εφαρμόζονται σε τελείως διαφορετικές καταστάσεις, ρεαλιστικός, πρακτικός προσανατολισμός και οδηγίες για τις ε, χώρες που έχουν προβλήματα με τα εργασιακά πρότυπα. Θα πρέπει να είναι και δυνατό, δυνατή προσαρμογή ε, στις διάφορες ανάγκες και διαφορετικές καταστάσεις επιτόπου. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ κυρία Σμίθ, λέει πρόεδρος. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Ζερόμ Σαπλιέ. Α, όχι, να αλλάξουμε. Την κυρία Μαριών Βερονίκα Αντιέ που είναι υπεύθυνη για τα προγράμματα ε, στο Γραφείο Παγκοσμιοποίηση και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων τη Διεθνή Ομοσπονδία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ για τη δυνατότητα να έρθω να μιλήσω. Είμαι πρόσωπος τη Διεθνή Ομοσπονδίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα ήθελα να πω κάποια πράγματα, να μοιραστώ κάποια απορίσματα των ερευνών μα όσον αφορά τι παραβιάσει που διαπιστώσαμε, όσον αφορά τα δικαιώματα των εργαζομένων. Αφήσαμε ένα-δύο αντίγραφα των εκθέσεων και θα αναφερθώ σε κάποιες ε, μελέτες. Θα επιλέξω παρόμοιες περιπτώσεις μαθές του κυρίου Μπένεντικτ. Αφού παρουσιάσω τις έρευνες θα καταλήξω στις στάσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με τα προβλήματα που εντοπίσαμε. Κάνουμε αποστολές σε εθνές επίπεδο, εξετάζουμε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο λιανεμπόριο σε παγκόσμιο επίπεδο στα πλαίσια συμφωνιών συνεργασίας με την Carrefour που είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος φορέας λιανικής στον κόσμο. Θέλουμε να βελτιώσουμε τις συνθήκες των εργαζομένων στην αλυσίδα εφοδιασμού και να εξασφαλίσουμε τα δικαιώματά τους γίνονται σεβαστά. Αυτή η συμφωνία συνεργασία επιτρέπει την αξιολόγηση παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην αλυσίδα εφοδιασμού με τη πρόσβαση στα διάφορα εργοστάσια όταν κάνουμε αποστολές, επίσης συναντώμεθα με την τοπική αυτοδιοίκηση, εθνική κυβέρνηση, μη κυβερνητικέ οργανώσεις, συνδικάτα, ε, ντόπιου παραγωγούς και ενώσεις ε, επιχειρήσεων και μετά κάνουμε συστάσεις και κάνουμε συστάσεις και συγκεκριμένα στο Καρφούρ και έχουμε, κάνει, έχουμε συντάξει εκθέσεις, έχουμε αντίγραφα εδώ για να τα πάρετε. Ερχόμαστε σε επαφή με επιχειρήσεις, ε, με τα κράτη εστιαστήκαμε για τις μελέτες μας στην ε, Ασία και στον τομέα της κλωστοϊφαντουργίας μέχρι τώρα. Ξεκινά από την Κίνα. Κάναμε αποστολή τον Νοέμβριο του 2012 στην επαρχία Γκουαντόγκ, στα νοτιοανατολικά της Κίνας. Και τι διαπιστώσαμε επισκεπτόμενοι διάφορα εργοστάσια παράγουν προϊόντα γνωστά ότι υπάρχουν παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των εργαζομένων μάλλον, κυρίως όσον αφορά τις υπεργολαβίες και όσον αφορά τους εισαγωγείς. Υπάρχει έλλειψη διαφάνειας. Υπήρχε πλήρης έλλειψη ελευθερίας ε, συνεταιρίζεστε, συλλογικών διαπραγματεύσεων, κοινωνικού διαλόγου. Υπήρχαν προβλήματα μεγάλο υπερορία 40 ώρες εργασίας την εβδομάδα προβλέπονται στην Κίνα. Οι περισσότεροι εργαζομένοι όμως πήγαιναν 60 και 80 ώρες την εβδομάδα και είδαμε και επισφαλή συνθήκες εργασία, χαμηλές αμοιβέ χαμηλά ομολομίστια καμιά φορά πληρώνονται με το κομμάτι εργαζόμενοι, έτσι εξηγούνται και οι υπερορίε. Σε κάποιε περιπτώσει οι εργαζόμενοι δεν είχαν συμβάσει εργασία και παρά το ότι το κινέζικο δίκαιο προβλέπει κάτι τέτοιο, δεν, ε, και ήταν δυνατότητα επιλογή, δεν ήταν υποχρεωτική περίθαλψη. Μετά με, συντάξαμε την Ινδία, Ιούλιο 2013 Πήγαμε σε αποστολή, πήγαμε στην Ινδία, επισκεφτήκαμε διάφορα εργοστάσια σε τρεις πολιτείες, Τέμερατζούς, Ούτρα και Χαριάνα. Και βρήκαμε ότι ε, υπήρχαν σημαντικές παραβιάσεις ε, των συμβάσεων του, της Διεθνούς Οργανώσης Εργασίας και είδαμε και το πρόγραμμα του Σουμαγκάλι που είναι ένα πρόγραμμα προσλήψεων όπου νέα κορίτσια προσλαμβάνονται κυρίως από την Ήπεθρο και πάνω και εργάζονται σε διάφορα εφαντουργία ε, και έχουν συμβάσεις ε, ορισμένου χρόνου και μετά τους δίνεται ένα αποκοπήν ποσό για την πρίκα τους. Αλλά οι συνθήκες ήταν ε, πάρα πολύ κακές τελικά. Λοιπόν, σε διάφορα εργοστάσια ενδύσεως υπήρχαν ελλείψεις συνδικάτων στην Ινδία και υπήρχαν και πρακτικά εμπόδια όσον αφορά την κατάρτιση, τη διαμόρφωση μάλλον συνδικάτων. Υπήρχαν και άλλοι παράγοντες αρνητικοί, συνθήκες εργασίας, ε, επισφαλείς συνθήκες εργασίας, όσον αφορά τις συνθήκες μαθητείας δεν ήταν καλές, τα μορομίστια ήταν πάρα πολύ χαμηλά, υπήρχαν θέματα διακρίσεων κατά των μεταναστών και διαφορές λόγω του φύλου. Ε, εντάχει τώρα Μπαγκλαντές που ανέφερε και ο συνάδελφος η αποστολή έγινε το 2007 και τότε διαπιστώσαμε ότι δεν υπήρχε ελευθερία του συνεταιρίζεστε, δεν υπήρχε παρκέ ημερομίσθιο, δεν υπήρχε κάλυψη, δεν υπήρχε πρόγραμμα επίλυση διαφορών, πρόβλημα ε, με τι υπερορίε. Είδαμε την τραγωδία που έγινε στο Ράνα Πλάζα και ξέρουμε ότι υπάρχουν ακόμα ανησυχίε για τι συνθήκε εργασία, θέματα ασφαλεία, ε, αποζημίωση κλπ. Υπάρχουν προβλήματα όσον αφορά τι επιθέσει, κατά των ηγετών των συνδικάτων. Εκδώσαμε έκθεση σχετική το 2013 που αναφέρει συγκεκριμένα για τις, στις επιθέσεις κατά των επικεφαλής των συνδικάτων. Ο Αμινούλ Ισλάμ δέχθηκε επίθεση και σκοτώθηκε και δεν εξηχνιάστηκε ο θάνατός του. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε επίσης ότι υπάρχουν ανθρώπινα προβλήματα σε εργοστάσια και στην Ευρώπη, στην Ισπανία όπως στις καλλιέργειες φράουλα στην Ισπανία υπάρχει διεθνής διάσταση του προβλήματος. Το εργατικό δυναμικό βασικά αποτελείται από μαροκινούς, εργαζομένους, μετανάστριες που έρχονται εποχιακά. Παρόμοια προβλήματα είδαμε σε εργοστάσια και στην Ευρώπη. Συγκεκριμένα όσον αφορά την πρόσβαση στα συνδικάτα, δεν υπήρχε πρόσβαση στα συνδικάτα για προσωρινούς εργαζομένους, θέματα διάκρισης, δεν καλύπτεται ούτε καν το ελάχιστο εισόδημα παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων λοιπόν ε, διαρκούν και θέλω να τονίσω ότι αυτή τη στιγμή οι παραβιάσεις γίνονται και κατόπιν και πιέσεων πασκούνται ασκούνται στους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ε, αλληλένδετα είναι τα προβλήματα. Βλέπουμε μέσω της έρευνας ότι οι υπερασπιστές, οι υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων καταγγέλουν επιχειρήσεις και είναι θύματα επιθέσεων και παρενόχλησης νομικής βιοπραγιών και καμιά φορά φτάνουν και σε φόνο. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα ρόλο να παίξει σχετικά με τα προβλήματα αυτά, όπω οι κατευθύνση γραμμή τη Ευρωπαϊκή Ένωση για του προσπιστέ των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Συνάδελφο αναφέρθηκε στο παράδειγμα τη Καμπότζη, όπου εργαζόμενοι στον τομέα τη ένδυση ζητούσαν ένα ημερομίσθιο επαρκέ για να επιβιώσουν και πυροβόλησαν πραγματικά πειρά στα πλήθη. Φυλακίστηκαν πολλοί επιμακρών, πολλοί τραυματίστηκαν και Κάποιοι σκοτώθηκαν κιόλα. Τα, στα πορίσματά μας ε, βασιζόμαστε για συστάσεις. Οι εθνικές κυβερνήσεις τα λαμβάνουν αυτά και οι κατασκευαστές κάνουμε συστάσεις επιχειρήσεις. Γνωστές επιχειρήσεις σύμφωνα με τα πλαίσια του ΟΗΕ. Θέλουμε να σέβονται ανθρώπινα δικαιώματα να φροντίζουν στα του εργαζομένου. Οι πρακτικέ που εφαρμόζουν για τι αγορέ του να μην είναι τα δικαιώματα, χρειάζεται βελτίωση διαφάνεια, χρειάζεται να πιεστούν οι προμηθευτέ για τη βελτίωση συνθήκων εργασία και να πιεστούν και οι κυβερνήσει όπου αυτό ενδείκνυται. Τι διαπιστώνουμε όταν κάνουμε συστάσει στι επιχειρήσει, ότι εθελοντικοί ιδεολογικοί κώδικε και διάφορες μέθοδοι που χρησιμοποιούνται δεν επαρκούν για να αποφύγουμε σοβαρέ παραβιάσεις των δικαιωμάτων στην αλυσίδα εφοδιασμού. Όπως στην Ινδία υπάρχουν σοβαρά προβλήματα. Πήγαμε στα εργοστάσια και είδαμε ότι εκεί οι βιομηχανίες είχαν συνηθίσει να έρχονται οι ξένοι ε, αγοραστές να κάνουν ελέγχους και προσπαθούσαν να δείξουν ότι είναι ιδιώδεις συνθήκες, προσαρμοζόταν άμεσα. Και ήταν ανέφικτο για εμά να αξιολογήσουμε τι πραγματικέ συνθήκε εργασία. Διότι οι εργαζόμενοι δεν ήταν ελεύθεροι να μιλήσουν, του πίεζαν. Υπάρχει κάλυψη κυρίως όσον αφορά την ελευθερία του συνεταιρίζεστε. Σε κάποια εργοστάσια υπάρχουν επιτροπές εργαζομένων, αλλά διορίζονται από τη δίκηση αυτή. Οπότε αυτό δεν αποτελεί επαρκή βήματα συζητήσεων για την ελευθερία του συνεταιρίζεστε. Λαμβάνοντας αυτά υπόψη τι λέμε. Λέμε ότι υπάρχει ανάγκη για ρύθμιση, για νομοθεσία, να επιβάλλονται υποχρεώσεις. Αυτές οι υποχρεώσεις όμως αποτελούν τμήμα των υποχρεώσεων των κρατών να προστατεύσουν του ανθρώπου από την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που προκαλούνται από τίτα μέρη. Οι εταιρείε έχουν υποχρέωση σε τα ανθρωπίνα δικαιώματα και οι χώρε θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι αυτό γίνεται. Υπάρχουν καθηγητέ γραμμέ του ΟΗΕ για τα ανθρωπίνα δικαιώματα, εφαρμόζονται εθελοντικά, αλλά ε, δηλώνουν εκ νέου τι υφιστάμενε υποχρεώσει τη κρατικέ για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά παραβιάσεων από τα μέρη συμπεριλαμβανομένων και των πολυεθνικών εταιριών και νομίζω ότι είναι σημαντικό να τονίσουμε και να ξεπεράσουμε τη συζήτηση αυτή η εθελοντική έναντι υποχρεωτική, εφαρ... εφαρμογή των μέτρων, διότι είναι υποχρεωμένα τα κάτι να θεσπίζουν νομοθεσία και να την εφαρμόζουν για τη συμπεριφορά των εταιριών. Μάλιστα, όταν αναφερόμαστε στην προστασία των πέντε δικαιωμάτων, υπάρχει ανάγκη ενός εφιούς κράματος εθελοντικών μέσων και υποχρεωτικών τέτοιων αλλά τα ρυθμιστικά μέτρα, τα υποχρεωτικά συμπεριλαμβάνονται. Θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται σε κάθε διάλογο με τι επιχειρήσει. Τι διαπιστώνουμε όμω, ότι κάποιοι λένε ότι οι ρυθμίσει χρειάζονται ούτω ώστε να υπάρχει διεθνέ πλαίσιο ισότιμο. το, η Καρφούρ προσεκλήθη στον ΟΗΕ και τοποθετήθηκε η Καρφούρ και είπε ότι πρέπει να εφαρμόσει διεθνεί προδιαγραφέ. Σε κάποιε περιπτώσει οι επιχειρήσει ενθαρρύνουν αυτή την προσέγγιση. Λοιπόν, οι χώρες που φιλοξενούν πολυεθνικές εταιρείες όπως την Ευρώπη πρέπει να εφαρμόζουν νομοθεσία που απαιτεί επιχειρήσεις καταρχάν υποχρεωτικά να εφαρμόζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα για τις επιχειρήσεις τους και για τις σχέσεις με άλλες εταιρείε. με θυγατρικές κλπ. να εφαρμόζονται σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού οι χώρε υποδοχέ πρέπει να θαρρύνουν, να απαιτούν μεγαλύτερη διαφάνεια επιχειρήσει, να αποκαλύπτουν πληροφορίε για την αισίδα εφοδιασμού, για το πώ διαμορφώνεται η διοίκηση, ποιε είναι οι δραστηριότητε σε παγκόσμιο επίπεδο, ποια μέτρα λαμβάνονται για να ε, προστατεύονται οι εργαζομένοι. Θα πρέπει να υπάρχουν αποζημιώσει για θύματα παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σχετιζομένων με την εταιρεία, όπω και θύματα παραβιάσεων που είναι σε τρίτε χώρε, στο εξωτερικό. Να αποζημιώνται και αυτοί. Τι πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να καλύψει αυτά τα προβλήματα όταν υπάρχουν παραβιάσει που προανέφερα. Πρέπει να εξασφαλίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι τα κράτη-μέλη εφαρμόζουν τα αναγκαία νομοθετικά μέτρα. Επίση, να πιεστούν και οι χώρε και η Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτω ώστε να εφαρμόζεται στεναρό πλαίσιο σχέδιο δράση για την εφαρμογή το κατευθυντήριο γραμμών του ΟΗΕ για τις επιχειρήσεις ανθρώπινα δικαιώματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εξασφαλίσει το ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαδραματίζει έναν ενεργό ρόλο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι αρμόδιες γενικές διευθύνσεις θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξασφαλίζει συνοχή πολιτικών όσον αφορά τις εμπορικές διαπραγματεύσεις, σε διμερείς συμφωνίες που στο τέλος επηρεάζουν τα δικαιώματα των εργαζομένων στο εξωτερικό και έχουμε κινητοποιηθεί σαν φορέα στο θέμα αυτό. Ακολουθούμε, παρακολουθούμε τις διαπραγματεύσεις ελευθέρω εμπορίου με Λάος, Βιετνάμ και Αιγύπτο και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εξασφαλίσει συνοχή πολιτική όσον αφορά τι υποχρεώσει που έχει αναλάβει όσον αφορά του προασπιστέ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπω προαναφέρθηκε. Τέλο, πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συμμετέχει καλή την πίστη και πλήρω στη διαδικασία ανάπτυξη συνθήκων που ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2014 στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που προβλέπει τη δημιουργία δικυβερνητικής ομάδας εργασίας για τις επιχειρήσεις και ανθρώπινα δικαιώματα με εντολή να καταρτήσει νομικό μέσο για τις επιχειρήσεις ανθρώπινα δικαιώματα. Και πιστεύουμε ότι αυτό το μέσο είναι συμπληρωματικό. Συμπληρώνει περιφερειακές προσπάθειες και εθνικές τέτοιες για την ενίσχυση τη νομοθεσία και την επιβολή νομοθεσία. Οπότε η δικασία ανάπτυξη συνθήκη κατά τη συνθήκη και εφαρμογή τη κατευθυντήρια γραμμή του ΟΗΕ και τα εθνικά προγράμματα δράση πράγματι είναι συμπληρωματικά μεταξύ του και είναι βασικά ούτω ώστε να υπάρχει ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού για τι διεθνεί επιχειρήσει. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Ζερόμ Σαπλιέ, συντονιστή του Ευρωπαϊκού Συνασπισμού για την Εταιρική δικαιοσύνη. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε που μας δίνετε την ευκαιρία ανταλλαγής απόψεων με τα μέλη της υποεπιτροπής σας σε σχέση με την ευρωπαϊκή δράση για τις σε σχέση με τις επιχειρήσεις επιβεβαιώνω το ενδιαφέρον στο θέμα αυτό να συνεχιστεί η δουλειά και να δοθεί ακόμη μεγαλύτερη σημασία όπως υπογραμμίστηκε και κατά τη διάρκεια της προηγουμένης θητείας από την υποεπιτροπή σας. Θα ήθελα να αναφερθώ τώρα σε μια συμμαχία με 11 πλατφόρμες από 15 ε, με πλατφόρμες από 15 ευρωπαϊκά κράτη και δράσεις κοινωνίας των πολιτών και ιδιαίτερα θα ήθελα να αναφερθώ στις ε, ε, δράσεις του Γενικού Γραμματέα για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα και το βαθμό στον οποίο μπορούν τα ευρωπαϊκά κράτη και επιχειρήσεις να συμβάλλουν. Όπως υπόθηκε ήδη, παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων από τις επιχειρήσεις λαμβάνουν χώρα εκτός Ευρώπης σε χώρες που έχουν λοιπές ε, κράτος δικαίου, διαφθορά και ανεπαρκές δικαιοδοτικό σύστημα και επιπλέον μέσα σε αυτό το χαλαρό περιβάλλον, δεν υπάρχει υπεύθυνη συμπεριφορά των μητρικών εταιριών στις, ε, σε σχέση με τις ε, θηγατρικές τους ή τους εμπορικούς εταίρους. Έτσι λοιπόν προκύπτει όλο και περισσότερο, όλο και μεγαλύτερος αριθμός παραβιάσεων ανθρώπινων δικαιωμάτων και γενική ατιμορρησία. Οι διεθνείς διατάξεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα υποχρεώνουν τα κράτη-μέλη να, τα συμβαλόμενα μέρη να, προστατε, να αποτρέπουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, να και να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα ακόμη και όταν αυτά παρουσια, παραβιάζονται από κάποιου άλλου. Δηλαδή αυτό έχει σαν συνέπεια την εξουεδαφικότητα και καθημερινά λαμβάνονται αποφάσει σε έδρε επιχειρήσεων στο Παρίσι, το Λονδίνο, το Βερολίνο, τη Μαδρίτη που έχουν άμεση επίπτωση ω προ τι δράσει ε, θηγατρικών, υπεργολάβων, ε, προμηθευτών και ω εκ τούτου συνέπειε στη ζωή εκατομμυρίων και δισεκατομμυρίων εργαζομένων εκτό Ευρώπη. Οι αρχέ λοιπόν, λοιπόν κατευθυντήριες αρχές για τις αρχές των επιχειρήσεων που εκδόθηκαν, υπογραμμίστηκαν και υποστηρίχθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία υποσχέθηκε να τι ενσωματώσει σε μελλοντικέ τη δράσει, σαν κυρίαρχο κομμάτι τους. Και θα ήθελα πολύ σύντομα να παρουσιάσω μια επισκόπηση των δράσεων αυτών της Ευρωπαϊκής Ένωση και των κρατών Μαλών, ιδιαίτερα όμω να υπογραμμίσω δύο κύρια σημεία αυτών των ε, κατευθυντηρίων ε, αρχών των Ηνωμένων Αθηνών που δεν έχουν υπογραμμιστεί επαρκώ. Καταρχάς την ανάγκη κεντρική έννοια της ε, ε, λογικής επιμέλειας ε, της αρμόσας επιμέλειας και η δυνατότητα για την δικαστική προσφυγή. Όσον αφορά την ε, λογική ή αναμενόμενη επιμέλεια, οι Ηνωμένες, τα Ηνωμένα Έθνη καλούν τα κράτη-μέλη να ε, υλοποιήσουν αυτή την αρχή, δηλαδή να εντοπίζουν, να προλαμβάνουν και να αποκαθιστούν τέτοιου είδους παραβιάσεις. Αυτό αφορά όλες τις επιχειρήσεις συμπεριλαμβανομένων και των θηγατρικών και των εμπορικών εταίρων τους. Αυτό αυτή η αρχή του due diligence έχει το δυναμικό πιστεύουμε να επηρεάσει την ε, συμπεριφορά μιας, ενός μεγάλου αριθμού επιχειρήσεων και να οδηγήσει σημαντικές αλλαγές. Σε παραδείγματι, αν οι κύριοι Λιανοπολιτές απαιτούσαν πάντοτε να υπάρχει εκπροσώπηση των εργαζομένων στις ε, επιχειρήσεις από τις οποίες προμηθεύονται τα προϊόντα τους, θα είχαμε σημαντική αλλαγή. Επίσης, αν είχαμε πιο, σοβαρό, πιο μεγάλη σοβαρότητα στην κοινωνική ευθύνη των επιχείρησεων της Ευρώπης ε, μέσα από ένα νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο όμως δυστυχώς ακόμη δεν έχει υλοποιηθεί και έχει βρίσκεται μόνο σε θελοντική βάση, θα μπορούσε, όπως απέδειξε μια διεθνής μελέτη, να ε, οδηγήσει αυτό το due diligence ε, σε τομείς συναφής με τα ανθρώπινα δικαιώματα, διαφθορά, ασφαλή στον χώρο εργασία περιβάλλον, σε σημαντικές αλλαγές και πιστεύουμε ότι θα έπρεπε, για να μην είναι μόνο μπορούσε, να είναι και εκτιμένο στα δικαιώματα των εργαζομένων για όλες τις επιχειρήσεις. Επειδή θέλω να αναφερθώ στην πρόσβαση στη δικαιοσύνη, τη δυνατότητα δηλαδή για προσφυγή και ουσιαστική αποκατάσταση ζημίας για το θύμα, όπως άλλωστε περιγράφεται και στις κατευθυντήριες ε, αρχές των ΗΕ, αλλά που δεν έχει κοινοποιηθεί επαρκώς σε επίπεδο ούτε Ευρώπης. Μηχανισμός εξοδικαστικός λοιπόν καταρχάς επίλυσης διαφορών, διαμεσολάβηση μεταξύ επιχειρήσεων, σημεία επαφή σε πλαίσιο όσα, χρήσιμοι μηχανισμοί που όμως θα πρέπει να αποδειχθούν πιο αποτελεσματικοί, γιατί είναι πολύ λίγοι αυτοί που σήμερα έχουν μια αποτελεσματική πρόσβαση στην ε, δικαστική, στην ε, διευθέτηση των διαφορών, η οποία όμως διαφορών δεν μπορεί να υποκαταστήσει την πρόσβαση στα δικαστήρια, ανεξάρτητα δικαστήρια, για να δίνεται μια ουσιαστική λύση στα προβλήματα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν εμπόδια όμω οικονομικά, δημοσιονομικά, ε, δικονομικά, τα οποία καθιστούν αδύνατη σχεδόν την προσφυγή ενό εργαζομένου θύματο ε, μιας άρνησης παροχής ε, δικαίωσης στην πατρίδα του σε δικαστήρια της Ευρώπης. Ελάχιστες είναι οι δίκες οι οποίες έχουν καταλήξει τιμιγορίες στο Ηνωμένο Βασίλειο της κατοχώρας και κανένα που βρίσκονται ακόμη εν εξελίξει στη Γαλλία είχε η Ευρώπη τα τελευταία χρόνια δείξει απροθυμία για δέσμευση της δικαιοσύνης της ε, σε θέματα που έχουν να κάνουν με τις διεθνείς δραστηριότητες των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Πρέπει ιδιαίτερα να υπογραμμίσουμε ότι τα εμπόδια που καταγράφονται στα ανθρώπινα δικαιώματα συσχετίζονται και με άλλα αντίστοιχα για την προστασία των καταναλωτών, την προστασία, του περιβάλλοντος κτλ. Και θεωρούμε ότι είναι πρωταρχική σημασία η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη της να εξετάσουν τα εμπόδια αυτά ως προς την πρόσβαση στη δικαιοσύνη και να τα, να τα καταρρύψουν. Ε, θα ήθελα επίσης να πω ότι σε ένα έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με το Czech Frank Bold ε, ε, πρόκειται να οργανωθεί στις 12 Νοεμβρίου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μια δέσκευση υψηλού επίπεδου με, αντικείμενο συστάσεις για πραγματικά ηγετική θέση στο θέμα αυτών των δικαιωμάτων. Επίσης ήθελα να αναφερθώ στις κατευθυντήριες γραμμές ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2011 έχουν αναλάβει προσπάθειες και τα κράτη-μέλη για να υλοποιήσουν τις δεσμεύσεις σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις επιχειρήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Για να κοιταχτούμε λίγο στον καθρέφτη θα έλεγα ότι έχουμε μια πολύ ε, διστακτική προόδο. Οι κατευθυντήριες αρχές έχουν ενσωματωθεί σε ένα βαθμό με την ανακοίνωση του 2011 για τις επιχειρήσεις η οποία ανακοίνωσε ισχύει το 2014 και η οποία προβλέπει δέσμευση για την ανάπτυξη ενό σχεδίου σχεδίου με προτεραιότητε για την υλοποίηση των κατευθυντήριων αρχών που θα πρέπει να ακολουθηθεί και από αντίστοιχε δράσει των κρατών μελών. Αυτό το σχέδιο ακόμη ε, έρχεται, δεν έχει ακόμη παρουσιαστεί. Τρία κράτη μόνο έχουν παρουσιάσει εθνικά προγράμματα δράση. Οι κατευθυντήριε αρχέ λοιπόν και η αρχή του due diligence ε, καταγράφονται και αντικατοπτρίζονται σε κάποιε ευρωπαϊκέ ε, μεταρρυθμίσει που είναι εν εξελίξη, έχουν ολοκληρωθεί. Παραδείγματι, πρόταση κανονισμού για το εμπόριο ορυκτών προερχομένων από, ε, ένοπλες, ε, από ε, εμπόλεμες περιοχές, το οποίο όμως βρίσκεται σε εκούσια βάση και δεν είναι υποχρεωτικό. Τον Απρίλιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, εξέδωσε μια απόφαση για την μη οικονομική λογοδοσία των επιχειρήσεων. Είναι αρκετές οι επιχειρήσεις οι οποίες ε, είναι υποχρεωμένες να δώσουν λόγο για τις συνέπειες της δράσεώς τους ως προς το περιβάλλον αλλά και τα εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι κάποιο σημαντικό βήμα ασφαλώς αλλά δεν είναι υποχρεωμένες παρότι υπάρχει το due diligence ε, δεν είναι υποχρεωμένε οι επιχειρήσει να εφαρμόσουν την αρχή του due diligence. Δηλαδή, μπορούν να κάνουν μια ανακοίνωση που θα λέει ότι δεν έχουν, δεν έχουν μέσα ώστε να εφαρμόσουν το due diligence. Και επίση θα ήθελα να αναφερθώ στη μεταρρύθμιση τη οδηγία για τι δημόσιε προμήθειε, η οποία δεν επέτρεψε την ε, πρόοδο που θέλαμε ε, σε σχέση με τα είναι εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τι επιχειρήσει και, και την τήρηση των κατευθυντηριών αρχών. Ε, υπάρχουν κάποια μέσα καθοδήγησης, ε, οδηγία, εγχειρίδια για τις επιχειρήσεις και ένα εγχειρίδιο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δίνουν κάποιες συστάσεις μόνο. Θα ήθελα λοιπόν ε, να καταλήξω σε ένα μήνυμα το οποίο είναι κατεπήγον πλέον να αναλυφθεί ε, στρατηγική σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Χρειάζεται μια στρατηγική και ένα σχεδιασμός στεναρός. Αυτή τη στιγμή απουσιάζουν. Τρεις διαδικασίες είναι εξελίξη, τρεις διαδικασίες οι οποίες μπορούν να προσφέρουν τη δυνατότητα να θέσουμε τα ορόσημα μια στρατηγική τέτοιου τύπου και τις ανέφερα νωρίτερα. Εδώ έχουμε να κάνουμε λοιπόν με το σχέδιο που αναμένεται να κατευθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την υλοποίηση των κατευθυντηρίων αρχών ε, δεν υπήρξε η πολιτική βούληση ή ηγετική πρωτοβουλία στο επίπεδο αυτό, αλλά χάρη στις ε, πιέσεις τη Γενική Διεύθυνση για των Επιχειρήσεων έχουμε μια σημαντική ε, στελέχωση από τι γενικέ διευθύνσει απασχόλησης κοινωνικών θεμάτων, εξωτερική δικαιοσύνη και άλλων θεμάτων ε, και άλλων αρμοδιοτήτων που βλέπω εδώ παρόντες ε, εκπροσώπου του σήμερα έχουν ε, προχωρήσει σε μια συνεργασία αλλά δεν έχουμε σε ανώτατο επίπεδο τη δέσμευση που θα μα επέτρεπε να δούμε μια εγκάρσια στρατηγική σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μια άλλη δυνατότητα για ορόσημα ω προ τα δικαιώματα αυτά και το σεβασμό του από τι επιχειρήσει είναι το θέμα τη εταιρική ευθύνη και τη στάση την οποία θα πρέπει να τηρήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ορίσει ε, να θέσει το ύψος των φιλοδοξιών σε σχέση με την ευθύνη που θα δείχνουν οι επιχειρήσεις ε, ως προς την κοινωνία στην οποία δραστηριοποιούνται. Μια άλλη δυνατότητα, ένα στρατηγικό πλαίσιο που πρόκειται να υιοθετηθεί του χρόνου και θα πρέπει να περιλαμβάνει κεφάλαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων και επιχειρήσεων. Επομένω, ναι, τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι επιχειρήσεις ενσωματώνονται όλο και περισσότερο στι ε, υπηρεσίε, σαν έννοια, είναι όλο και πιο εγκάρσια η θεώρηση, το βλέπουμε και στην δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά συνέπεια απόλυτη δεν υπάρχει. Είναι ασθενεί ακόμη οι κινήσει. Ε, οι εμπορικέ πολιτικέ ε, που έχουν συνέπειε στα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων έξω από την Ευρώπη δεν έχουν ακόμη προχωρήσει. Μιλάμε για ένα ευφυέ μείγμα, smart mix, μιλάμε για εθελοντικέ προσεγγίσει, επομένω μόνο ευσεβεί πόθου και δεν έχουμε δει καμία σαφή βούληση για τη θέσπιση υψηλού επίπεδου προδιαγραφών για τι επιχειρήσει Μόνο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με την υποεπιτροπή σα μπορεί να καθοδηγήσει ε, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ε, πορεία αυτή και τη δέσμευση. Γι' αυτό λοιπόν το μήνυμα που θέλω να σας δώσω είναι ένα μήνυμα ε, αισιοδοξία και ενθάρρυνση να συνεχίσετε να πιέζετε. Σε επίπεδο διεθνέ έχουν προχωρήσει κάποια ζητήματα ε, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Δανία, οι κάτω χώρε έχουν προχωρήσει με εθνικά σχέδια, η Ισπανία, η Ιταλία, η Φιλανδία έχουν προχωρήσει αρκετά. Κάποια κράτη δείχνουν ότι σκοπεύουν να δημοσιεύσουν τα σχετικά του σχέδια, αλλά τα περισσότερα από τα σχέδια που ε, δημοσιεύονται δυστυχώς δείχνουν μόνο ε, προθέσεις για εθελοντικές δεσμεύσεις και δυστυχώς δεν περιλαμβάνουν καμία δεσμευτική ε, υπαγωγή στην εθνική δικαιοσύνη. Το δε σχέδιο της Δανίας έχει καθαρά έξω, ε, ένδο εδαφικό χαρακτήρα. Για τη Γαλλία ένα σχέδιο νόμου βρίσκεται υπό Σχέδιο νόμου που αφορά την υποχρέωση επιμέλειας της μητρικής εταιρείας σε περίπτωση παραβίασης θεμελιωδών δικαιωμάτων από τις θηγατρικές, κάτι το οποίο παρακολουθούν αρκετά κράτη-μέλη πιστεύω με ενδιαφέρον. Το Ρεμένο Βασίλειο εκδίδει ένα σχέδιο, έχει επεξεργαστεί ένα σχέδιο νόμου για τη σύγχρονη δουλεία ε, εν γέννη βλέπουμε ότι λίγα είναι τα κράτη-μέλη τα οποία είναι διατεθειμένα να εισαγάγουν τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις. Χρειάζεται μια συντονισμένη προσέγγιση, την οποία δεν έχουν αυτά τα κράτη-μέλη ακόμα και ίσως αυτό να αποτελεί μια ε, βολική αλλά πάντω ανεπαρκή δικαιολογία και θα πρέπει να αισθανθούν να συνεχίσουν τι μεταρρυθμίσει και σε εσωτερικό επίπεδο. Άρα πιστεύουμε ότι είναι πολύ κατακαιρματισμένη η προσέγγιση, δεν υπάρχει στρατηγική, δεν υπάρχει φιλοδοξία, δεν υπάρχει ηγετική θέση. Από το 2008 και αυτά είναι στοιχεία τη ε, εταιρεία Mavercraft, ανάλυση κινδύνου, αύξηση άνευ προηγουμένου 70% παραβιάσεων των ανθρώπινων δικαιωμάτων ανά τον κόσμο και είναι στιγμή πλέον με την αυτή νομοθεσία Ευρωπαϊκή Ένωση να επιδείξει φιλοδοξία να αναγνωρίσει τη σημασία, την έκταση του προβλήματος, να εντοπίσει τις απαραίτητες νομοθεσίες, να εισαγάγει μια στρατηγική εγκάρσια με βάση τις κατευθυντήρες αρχέ των ΗΕ και ιδιαίτερα όσον αφορά την εύλογη επιμέλεια και τη δυνατότητα πρόσβαση της δικαιοσύνη, στη δικαιοσύνη σε, θέμα, ε, σε θέματα αστικού αλλά και ποινικού δικαίου και βεβαίως θα πρέπει να ε, παρακολουθήσει τις ε, συστάσεις του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών. Η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν είναι απλώς μια ωραία ιδέα, είναι μια απέτηση με την οποία βρίσκεται καθημερινά αντιμέτωπος ο νομοθέτης προκειμένου να προστατέψει τον εργαζόμενο, είτε αυτός βρίσκεται στη γωνία του δρόμου, είτε βρίσκεται και εργάζεται σε ένα εργαστήρι στο Μπαγκλαντές. Ευχαριστώ. Και... Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Σαπλή. Θα δώσω τώρα το λόγο στα μέλη της Επιτροπής μας και εν συνεχεία μπορείτε και εσείς εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης να τοποθετηθείτε. Όπως βλέπετε, έχουμε να κάνουμε με ένα ευρύτατο πεδίο παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ουσιαστικά δεν υπάρχουν νομικά μέσα, τόσο σε διεθνές ε, όσο και σε εθνικό επίπεδο, για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού. Είναι προφανές ότι η παγκοσμιοποίηση των αγορών δεν συνοδεύτηκε και με παγκοσμιοποίηση των δικαιωμάτων. Επίσης προφανές είναι ότι το ζήτημα είναι ιδιαίτερος λεπτό στις κοινωνίες μας, στις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό στην υποεπιτροπή μας να τονίσουμε και να ε, ασκήσουμε αν θέλετε και πίεση και για την ευαισθητοποίηση και πληροφόρηση της ευρωπαϊκής κοινής γνώμης που πολλές φορές δεν έχει στη διάθεσή της πληροφορίες και δεδομένα για το θέμα αυτό και βέβαια θα πρέπει ταυτόχρονα να προωθήσουμε και τη διεθνή νομοθεσία και την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Τόσο λεπτό είναι το θέμα, ώστε τώρα που δεν μας ακούει κανείς, μπορώ να σας πω ότι ήταν λεπτό ακόμη και το ότι εμείς θελήσαμε να θέσουμε το ζήτημα ε, στην Μέσια Διάταξη και να το συζητήσουμε. Άλλες επιτροπές που δραστηριοποιούνται σε άλλους τομείς ε, Πραγματικά το πλαίσιο του, μάλλον το περιεχόμενο της ακρόασης και το ότι συμπεριλάβαμε κάποιες, ε, μάλλον ζήλεψαν και έπρεπε να βάλουμε λέξεις μέσα στην ακρόαση ώστε να φαίνεται ότι περιλαμβάνουμε μόνο τα δικαιώματα των εργαζομένων και τα δικαιώματα σε τρίτες χώρες. Αυτό σημαίνει ότι ακριβώς αυτό που πρέπει να κάνει η Επιτροπή μας είναι να εμβαθύνει, ε, να φτάσει μέχρι το βυθό σε αυτό το θέμα. Βέβαια δεν θέλουμε ε, να μπουν σε δεύτερο πλάνο άλλε επιχειρήσει, αλλά σε πρώτο πλάνο να μπουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Άλλε, συγγνώμη, επιτροπέ. Θέλουμε να μπουν σε πρώτο πλάνο τα ανθρώπινα δικαιώματα και ο τρόπο με τον οποίο δραστηριοποιούνται σε τρίτε χώρε οι ευρωπαϊκέ επιχειρήσει, που είπατε ότι έχουν κέρδη παράγουν κέρδη μεν, αλλά πολλές φορές ε, στο βωμό ε, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της υγείας, ε, εργαζομένων, πολλές φορές ανηλίκων, πολλών γυναικών, που βιώνουν πραγματικά συνθήκες πραγματικής δουλείας. Και νομίζω ότι η Επιτροπή μας πρέπει να εργαστεί σε βάθος και μπορεί να υπάρχει επιφύλαξη από άλλες επιτροπές, αλλά εμείς δεν πρέπει να ε, το αφήσουμε αυτό να μας σταματήσει. Παρακαλώ, έχετε το λόγο, κύριε Λοχμπίλερ. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω γερμανικά. Και σας ευχαριστώ ιδιαίτερως για την ε, πρωτοβουλία να οργανώσετε αυτή την ακρόαση εδώ. Έχουμε αρκετό χρόνο ώστε να ακούσουμε αρκετές και διαφορετικές ε, παρεμβάσεις που θα είναι πάρα πολύ χρήσιμες για την προσεχή δουλειά μας την επόμενη πενταετία. Έχω αρκετές ερωτήσεις βέβαια συμπληρωματικές και επί τη ευκαιρία θα εκμεταλλευτώ τις γνώσεις των ε, ειδικών μας. Για εσάς από την ε, Διεθνή Οργανώση Εργασίας μας ε, παρουσιάσετε τη σύσταση να συμπεριλάβουμε το, το θέμα των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων στον διάλογο για τα εργασιακά δικαιώματα. Πολύ ωραίο αυτό. Αλλά εάν υπάρχει σωματείο συνδικαλιστικό σε μια χώρα που δουλεύει, που εργάζεται. Πολλές φορές ξέρουμε ότι σε ορισμένες χώρες βέβαια διώκονται τα σωματεία. Από την άλλη από... όμως ξέρουμε ότι υπάρχουν και κάποιοι οποίοι δραστηριοποιούνται υπέρ των δικαιωμάτων των εργαζομένων χωρίς να έχουν αυτή την ιδιότητα επισήμως αναγνωρισμένη. Έτσι λοιπόν ε, η Διεθνής Οργάνωση Εμπορίου, Εργασίας προσπαθεί να προστατεύσει αυτούς τους ε, αγωνιστές για τα δικαιώματα των εργαζομένων, οι οποίοι ενδεχομένως δεν μπορούν να ενταχθούν σε σωματεία ε, λόγω της νομοθεσίας της χώρας ή γιατί δεν γίνονται δεκτοί από το σωματείο. Για τον κύριο Μπένεντικτ. Αναφερθήκατε στη Βερμανία την Καμπότζη, ακούσαμε αρκετά λόγια για το Λάος και το Βιετνάμ, αλλά βέβαια υπάρχουν και οι διάφορες υποθέσεις της ε, Ταϊλάνδης και ιδιαίτερα από τον τομέα της Γαρίδας που παρουσιάζει χαρακτηριστικά ακόμη και καταναγκαστική εργασία. Θα ήθελα λοιπόν να μα δώσετε κάποιε πληροφορίε επιπλέον και ίσω είναι κάτι το οποίο μπορεί να κινήσει το ενδιαφέρον τη Επιτροπή Αλία, για να πούμε και τη φράση All About first. Και για τη Βερμανία κύριε Μπένεντεκτ. Έχουμε ήδη διατυπώσει επικρίσεις και εδώ απευθύνομαι και στην Επιτροπή Εξωτερικής Δράσης. Υπάρχει μια συμφωνία επενδύσεων διαπραγματεύση τώρα με τη Βυρμανία. Ε, εγώ λοιπόν βλέπω ότι η αξιολόγηση αυτή των ανθρωπινών δικαιωμάτων καθίσταται πάρα πολύ δύσκολη. Θέλω η, Επιτροπή, η Υπηρεσία Εξωτερικής δράση να μας εξηγήσει γιατί είναι τόσο δύσκολο να ασχοληθεί με το θέμα αυτό στη δουλειά τη, ενώ υπάρχουν τόσα πολλά και καλά παραδείγματα αλλού. Έχουμε ε, από την Ευρωπαϊκή Ένωση εγκρίνει το σύστημα γενικευμένων προφίλ ε, προτιμήσεων ε, χωρίς τη συμπερίληψη των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή τις κατάφορες παραβιάσεις όπως λέγαμε ε, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να αναλάβει ένα σύστημα, ε, να επεξεργαστεί ένα σύστημα παρακολούθησης των παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εμείς έχουμε ως ομάδα των πρασινών, μικρή ομάδα, ε, κάνει την πρόταση για δεσμευτικές αναφορές στη δουλειά αυτή που αναπτύσσουν ε, επιχειρήσεις ε, με έδρα την Ευρωπαϊκή Ένωση και μεταθέτουν τις δραστηριότητες τους εκτός Ένωσης. Δυστυχώς από τους ελιστές και από τους στηρητικούς δεν μπορέσαμε να βρούμε επαρκή υποστήριξη για την πρόταση μας αυτή, εξού και έμεινε κρεμής η πρόταση, αλλά ελπίζω στην επόμενη πενταετία να προχωρήσουμε καλύτερα. Για την κυρία Σμιθ. Ίσως έχετε και την επισκόπηση, εσείς συζητάμε πάντα στο Κοινοβούλιο πόσο καλό είναι οι επιχειρήσεις να ε, έχουν, είτε πρόκειται για διεθνούς δραστηριοποίηση επιχειρήσεις, είτε πρόκειται για επιχειρήσεις μέτρα την Ευρώπη, να ε, επιλέγουν την ε, αυτοδέσμευση και την, την δεοντολογία περισσότερο. Έχετε κάποια εικόνα για το πόσες είναι αυτές που τηρούν τους κανόνες δεοντολογίας και την αυτοδέσμευση. Ε, δεν μπορώ να ρωτήσω φυσικά για το ποιες είναι οι δικές σας προτιμήσεις, γιατί ήταν ξεκάθαρο αυτό που είπατε, ένα μείγμα και σαφείς ε, ρυθμίσεις είπατε ότι χρειαζόμαστε, αλλά για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλω να υποβάλω την εξή ερώτηση, γιατί βλέπω ότι ε, δεν τολμάει να διατυπώσει απαιτήσει για πιο αυστηρές προϋποθέσεις όταν πάμε στη Γενέβη για να συζητήσουμε με τους διπλωμάτες θέματα θέσπισης μιας ομάδας εργασίας που θα παρακολουθούσε ενεργητικά αυτά τα ζητήματα δεν εξασφαλίζουμε υποστήριξη. Η ερώτησή μου λοιπόν θα ήταν ποια είναι η θέση μας, η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης δηλαδή στις διαπραγματεύσεις αυτές και πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε δεσμευτικά μέσα. Για, κύριε, για σας κύριε Σαπέ και μπορεί να έχω καταλάβει λάθος αλλά ε, αναφερθήκατε στη δυνατότητα ενίσχυσης της προστασίας των θυμάτων δικαστικής προστασίας εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αναφερθήκατε και στα κράτη, στα εθνικά κράτη. Δεν είναι αυτό κάπως ε, δεν θα ήταν μια δυνατότητα να ρωτήσουμε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αν υπάρχει δυνατότητα για την προστασία των δικαιωμάτων των θυμάτων εκείνων επιχειρήσεων οι οποίε εδρεύοντα στην Ευρώπη έχουν εκτό Ευρώπη προξενήσει κάποια σημεία. Και με συγχωρείτε κύριε Πρόεδρε να διατυπώσω μια ακόμη ερώτηση γιατί και εσεί, ε, κύριε Σοπέ το αναφέρατε αυτό. Το είχαμε δει και σε μια προηγούμενη συνεδρία τη Επιτροπή μα, Μια μελέτη για τα δικαιώματα των ηθαγενών ε, πληθυσμών και τα ορυκτά από εμπόλεμες ζώνες. Είχατε εσείς λοιπόν αναφέρει ε, το ζήτημα ε, μιας διαδικασίας σε σχέση με την εξόριξη ορυκτών από τις εμπόλεμες περιοχές όπου θα μπορούσε η Επιτροπή μας να διεκδικήσει μια έκθεση για να δούμε τι, πώς ακριβώς στηρούνται τα ανθρώπινα δικαιώματα στις περιοχές αυτές. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας κύριε Λοχπίλερ και θα το ζητήσουμε. Κάνατε ερωτήσεις σχεδόν σε όλους ε, τους ε, παρεμβαίνοντες, αλλά έχετε και κάποιες ερωτήσεις προς την υπηρεσία εξωτερικής δράσης που θα ε, απαντήσουν στη συνέχεια. Να δώσω στους κυρίους Χούγκο Μπένετικ, Σμιθ και Σαπλιέ το λόγο. Εν συντομία παρακαλώ, γιατί υπάρχουν και άλλοι που έχουν στήσει το λόγο πλήν της κυρίας Λοχμπίλερ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Να απαντήσω εντάχει στην ερώτησή σας. Είναι σαφέστατο για μένα και για όλους μας τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα καθώς και τα δικαιώματα των εργαζομένων πηγαίνουν μαζί. Τα δικαιώματα των εργαζομένων θα μπορούσαν να είναι και ένα υποσύνολο του όλου προγράμματος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ελοχεύει ένας κίνδυνος που πρέπει να προσέξουμε σε κάποιες περιστάσεις όταν μιλάμε για ανθρώπινα δικαιώματα τίνουμε να σκεφτόμαστε δικαιώματα εκτός των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Γι' αυτό είναι σημαντικότατο να τονίζουμε τις δύο διαστάσεις. Τούτου λεχθέντος αναγνωρίζω ότι αν κάποιος ηγέτης σωματίου συλληφθεί, κάποιου συνδικάτου και αντιμετωπιστεί με τρόπο εντελώς αντίθετο με το διεθνές ή εθνικό δίκαιο αληθεύει επίσης ότι και άνθρωποι που δεν εργαζομένοι αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα. Έχουμε περιπτώσεις όμως όπου επικεφαλής συνδικάτου θα πολεμά για δικαιώματα ανθρώπων που ίσως να μην είναι εργαζόμενοι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να μιλάμε ταυτόχρονα για ανθρώπινα δικαιώματα καθώς και για τα δικαιώματα των εργαζομένων. Δεύτερη ερώτηση που απευθύνατε σε όλα τα μέλη του πάνελ από ό,τι κατάλαβα. Αν χρειαζόμαστε πολύ πιο δεσμευτικό μέσο, εργαλείο. Και αυτό συνδέεται με το σχόλιο του συναδέλφου εξεβονίμων της κυρίας Σμιθ. Να υπάρχει μια διεθνή σύμβαση που είναι πιο πρακτικά εφαρμόσιμη Πώς το εκλαμβάνω από τη θέση μου. Υποχρεωτικό, δεσμευτικό ότι όχι, αυτό είναι κάτι που δεν λύγει σαν θέμα. Το σημαντικότερο είναι η επιβολή ιουδήποτε νόμου. Αναφέρθηκε το καθήκον προστασίας είναι πολύ εύκολο να σπρώξει κανείς το πρόβλημα στα χέρια της κυβέρνησης που έχει υποχρέωση να προστατεύει. Όλοι γνωρίζουν όμως ότι η πρωταρχική ευθύνη μιας κυβερνήσεως είναι να προστατεύει τους πολίτες της. Δεν είναι αυτό το θέμα. Πολύ συχνά το ζήτημα που τίθεται είναι η επιβολή του νόμου. Αν πάρουμε μία διάσταση της υποθέσεως του Μπαγκλαντές, μία διάσταση λέγω, οι άλλες διαστάσεις δείχνουν ότι μπορούσε να κάνει περισσότερα κυβέρνηση. Συμφωνώ με αυτά που είπαν άλλοι συνάδελφοι. Έχουμε μια χώρα, σαν την Μπαγκλαντέ. 130 εκατομμύρια κατοίκου έχει. Και έχουμε 60 επιθεωρητέ εργασίε για όλη τη χώρα. Μπορείτε να κατηγορήσετε την κυβέρνηση, να τη πείτε ότι έχετε υποχρέωση να προστατεύετε. Αλλά πρέπει να του βοηθήσουμε να αντιμετωπίσουν αυτό το θέμα που έθεσα. Γι' αυτό υπάρχει σχέση μεταξύ αυτού που συζητούμε και της αναπτυξιακής βοήθεια και του σχετικού προγράμματος για την αναπτυξιακή βοήθεια. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ, κύριε Μπένεντικτ. Εάν επιτρέπετε, στα γρήγορα, να προβώ ένα σχόλιο. Τα συνδικάτα στις περισσότερες χώρες δεν κάνουν απαραίτητα τη διάκριση μεταξύ ενεργών μελών του Συνδικάτου και Πρασπιστών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Σε πολλές χώρες υπάρχει ε, συνεργασία αυτό. Στην ETUC η FTA στέλνει μια αποστολή στη Λευκορωσία, π.χ. χάρη. Συνεργαζόμαστε με αυτούς, με αυτό το φορέα, ούτω ώστε να συνεργάζεται ο φορέας με τα συνδικάτα τα ντόπια. Αυτή η διάκριση δεν υπάρχει πάντα, δεν είναι πάντα σαφής και σίγουρα δεν είναι πάντα τέτοια η επιθυμία των συνδικάτων στις χώρες ή και στο παγκόσμιο προσκήνιο. Το μοντέλο τώρα των αλυσίδων εφοδιασμού. Παντού παρόμοιο είναι. Μπορούμε να αναφέρουμε διάφορες χώρες στην Αμερικανική Ήπειρο. Το πρόβλημα με τη γαρίδα στην Ταϊλάνδη είναι κατά κάποιο τρόπο εξίσου άσχημο ή χειρότερο από πολλά άλλα προβλήματα, σε σχέση με άλλα προβλήματα, αν το συγκρίνουμε. Χαίρομαι που το αναφέρατε. Εμπλέκονται πολλοί Βιρμανοί που το έσκασαν από τη Βιρμανία και καταλήγουν εργάζονται συνθήκες παρόμοιες ή χειρότερες από αυτές στην πατρίδα τους. πραγματικά καταναγκαστικής εργασίας και αφόρητων συνθήκων εργασίας. Ένα κομμάτι του προβλήματος και της πρόκλησης είναι να εντοπίσουμε στόχους. Υπεύθυνες επιχειρήσεις εκτός Ταϊλάνδης. Το πλεονέκτημα της κλωστοϊφαντουργίας ποιο είναι. Ότι τα προϊόντα πάνε σε εταιρείες και σε μάρκες που είναι εύκολα εντοπίσιμες και στην Ευρώπη και αλλού. Δεν σημαίνει βέβαια ότι το πρόβλημα είναι μικρότερο. Σημαίνει ότι είναι δυσκολότερο να αντιμετωπιστεί. Σχετικά με τη Βυρμανία, να πω απλώς ότι συμμερίζω με την απογοήτευσή σας. Δηλαδή ότι το Κοινοβούλιο εν γέννη δεν ενστερνίστηκε τις διάφορες προτάσεις για περισσότερο έλεγχο και λογοδοσία από πλευράς ευρωπαϊκών ε, επιχειρήσεων. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Σμιθ. Ευχαριστώ. Όσον αφορά το ερώτημά σας, πόσες εταιρείες αναλαμβάνουν εθελοντικές υποχρεώσεις. Αν ρωτάτε πόσες εταιρείες χρησιμοποιούν διεθνή πλαίσια ο σα κατευθείας γραμμές ή άλλα πλαίσια. Δεν έχω στοιχεία πρόχειρα. Υπάρχουν όμως στοιχεία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να έχει κάποια στοιχεία. Ίσως να υπάρχουν σε διεθνές επίπεδο. Αν αναφέρεστε στον αριθμό εταιριών που αναλαμβάνουν εθελοντικές υποχρεώσεις στο CSR, στο πλαίσιο αυτό, είναι δύσκολο σχεδόν αδύνατο να το καταλάβουμε. Να το δούμε μάλλον, συγγνώμη. Υπάρχουν κάποιες εταιρείε που κάνουν αυτό που θα θεωρούσαμε ευρωπαϊκό πλαίσιο, ίσως να μην το αποκαλούν έτσι, ίσως ε, οι μικρότερες εταιρείε και υπάρχουν στατιστικά στοιχεία από αυτού. Πόσες εταιρείε αναφέρουν στοιχεία για την υπεύθυνση επιφορά των επιχειρήσεων. Επειδή δεν υποβάλλεις αναφορά δεν σημαίνει ότι δεν λαμβάνει κάποια μέτρα όσον αφορά την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Μπορώ να έρθω σε επαφή μαζί σας, να δώσω στοιχεία για το διεθνές πλαίσιο. Αλλά γενικά είναι δύσκολη η στατιστική επισκόπηση. Υπάρχουν κάποιοι συμβουλοί, συμβουλευτικοί φορείς που προσπάθησαν να έχουν στατιστικά στοιχεία όσον αφορά την υποβολή αναφορών και ενημέρωση. Αλλά οι εταιρείε που αναλαμβάνουν εθελοντική δράση όσον αφορά την εταιρική ευθύνη είναι πολύ δύσκολο να σας δώσω στοιχεία εκτός αν μπορεί να με βοηθήσει από αυτού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ, κύριο Σαπελή. Για το πρώτο ερώτημα, σε σχέση με την πρόσβαση στη δικαιοσύνη, δεν υπάρχει μία και μόνη λύση που να είναι απλή και θα λύσει το πρόβλημα εξάπαντος. Πρέπει να αναλυθεί δράση σε διάφορα επίπεδα, εθνικό, ευρωπαϊκό, διεθνές οι ουσιαστικές αρμοδιότητες ό,τι αφορά την πρόσβαση στη δικαιοσύνη είναι σε εθνικό επίπεδο και γνωρίζουμε ότι πολλά κράτη-μέλη δεν ε, θέλουν και πολύ να τους παγορεύει κάποιος άλλος τον τρόπο με τον οποίο θα οργανώσουν ε, το δικαστικό του σύστημα. Όμως, νομίζω ότι εκεί εντοπίζεται το πρώτο επίπεδο δράσης. Υπάρχει ευρωπαϊκή αρμοδιότητα, πράγματι, συλλογικές ε, προσφυγές, είναι ένα θέμα, μπορεί να επανέλθει ε, στο προσκήνιο εναρμόνιση δικαιοδοτικών κανόνων επίσης στα κρατη και αυτό είναι μια σύντηση που θα επανέλθει με πρωτοβουλία της ΓΔ Δικαιοσύνη. Η περιφερειακή επιλογή που προτείνεται για ευρωπαϊκά δικαστήρια είναι ενδιαφέρουσα ως πρόταση. Δεν είμαι βέβαια ε, εμπειρογνώμων για αυτό το θέμα, αλλά νομίζω ότι τα δικαστήρια που υπάρχουν έχουν εντολή απέναντι σε κράτη, όχι όμως απέναντι στις επιχειρήσεις μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Άρα πρέπει πρώτα απ' όλα να αλλάξει το καθεστώς, ε, το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, του Διεθνού Σπινικού Δικαστηρίου, ώστε να είναι δυνατή η προσφυγή στη δικαιοσύνη κατά επιχειρήσεων. Είναι μια επιλογή μακρόπνοη και μακροπρόθεσμη που όμως αξίζει κατά την άποψή μου να μελετηθεί ως ενδεχόμενο και για τη δημιουργία ίσως και ενός Ευρωπαϊκού Ποινικού Δικαστηρίου. Σε ό,τι αφορά αυτά τα μεταλλεύματα που εξάγονται ή εξορίζονται σε χώρες που βρίσκονται σε εμπόλεμη κατάσταση. Πράγματι υπάρχει πρόβλημα, πρέπει και η δική σας υποεπιτροπή να δώσει την προοπτική των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, για τα θύματα σε αυτές τις εκμεταλλεύσεις. Πρόεδρος, θα δώσω το λόγο σε άλλα δύο μέλη της ε, Επιτροπής μας και έπειτα θα ακούσουμε την ε, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης καθότι μας πιέζει λίγο ο χρόνος, μέχρι τις 11 και 4 το πρέπει να έχουμε ολοκληρώσει και υπάρχει στη συνέχεια συνεδρία του Διευρωμένου προέδρου Παντσέρη και Παγάθα Ορθουντούα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας Ευχαριστώ και εγώ τους παρόντες, τους εμπειρογνώμονες. Στην ακρόαση έχω δύο πράγματα που θα ήθελα να αναφέρω που αφορούν όλους στην συζήτηση. Πιστεύω ότι είναι δυσκολότατο να διεξαχθεί αυτή η συζήτηση. Διότι πιστεύω ότι υπάρχει επίγνωση ότι σήμερα και στην Ευρώπη ε, η συζήτηση αυτή πάει κατά της ροής των πραγμάτων δηλαδή σε διάφορες χώρες, μειώνεται η προστασία, μειώνουν τα δικαιώματα, προσπαθώντας να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων προς τα έξω. Η τάση λοιπόν, πώς να το θέσουμε, είναι να νομισματοποιηθούν, να, να δοθεί χρειά χρήματος ε, στα δικαιώματα σε εμπορική λογική μπαίνουμε και μειώνονται οι προστασίες προς εργαζομένους. Εσείς ασχολείστε άμεσα με τα προβλήματα αυτά. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι δημιουργείται και μια σειρά διαιρέσεων και διχασμό που δύσκολο να ελεγχθούν. Εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει πόλωση ε, στον χώρο εργασίας μεταξύ εκείνων που προστατεύονται και εκείνων όχι. Εκείνων που προστατεύουν τα δικαιώματα και εκείνων που δεν προστατεύουν. Αυτή είναι μια διαίρεση. Και μετά έχουμε την εξωτερική διέρεση στο εναγορά εργασία στην παγκόσμια. Διότι οι εργαζόμενοι Ευρωπαίοι δεν ζουν αυτή την έλλειψη των δικαιωμάτων ως παράγοντα που απαιτεί μεγάλη μάχη. Το βλέπουν σαν στοιχείο ανταγωνισμού. Είναι πάρα πολύ δύσκολο στοιχείο. Ήθελα να τα πω αυτό. Πιστεύω ότι είναι δύσκολο να λυθούν τα προβλήματα στην Κίνα. Αλλά α θέσουμε ε, κάποια στοιχεία προ συζήτηση. Χρειάζεται μια πλατφόρμα, μια βάση για την καταπολέμηση των ανισοτήτων, διότι είναι από τα βασικά αίτια ανισότητα των δυσκολιών να εφαρμοστούν ε, τα δικαιώματα σε όλους τους εργαζομένους. Πρέπει τα δικαιώματα του εργαζομένου να είναι στο επίκεντρο των εμπορικών συμφωνιών με άλλε χώρε, ούτω ώστε να αποφευχθεί το αντίθετο. Δηλαδή η έλλειψη δικαιωμάτων σε κάποιε χώρε να μολύνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι να γίνει το αντίστροφο. Η Διατλαντική Συμφωνία μπορεί να αποτελέσει βασικό στοιχείο που θα μπορεί ε, να οδηγεί σε κάποια αλλαγή ταχύτητα όσον αφορά τα γεγονότα αυτά. Υπάρχουν οικονομικοί παράγοντες σημαντική πτυχή της εξωτερικής πολιτικής και θα πρέπει να γίνει κεντρικό σημείο. Τέλος, κατά την άποψή μας, αυτή η συζήτηση που γίνεται για λιτότητα και ανάπτυξη στην Ευρώπη είναι σημαντική και για έξω. Θα πρέπει να γίνει μια συνολική σφαιρική μάχη. Το λέω σε σένα, Πρόεδρε. Θα ήταν σκόπιμο από αυτά που άκουσα να προωθήσουμε εμείς μια πρωτοβουλία με δύο επιτροπές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οικονομική και κοινωνικών υποθέσεων. Οι δύο επιτροπές συμμετάσχουν. Διότι πιστεύω ότι η νομοθεσία που έχουμε μπροστά μας τα πέντε χρόνια, κυρίως όσον αφορά την Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων και Απασχόλησης, ε, είναι μάλλον υποτονική. Η όλη θητεία φαίνεται υποτονική και δεν βλέπω να υπάρχουν μεγάλοι στόχοι και προπτικές για αυτήν την Επιτροπή. Ίσως στην ημερήσια διάταξη θα έπρεπε να μπουν ε, κάποια σημεία που είναι σημαντικά. Και κάτι άλλο. Ο ρόλο των, ευρωπαϊκών επιχειρήσεων εκτό Ευρωπαϊκής Ενώσεω, Εκεί που τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν γίνονται σεβαστά. Η κυρία Κατιά αναφέρθηκε σε αυτή την ομάδα, τη διακυβερνητική για την εργασία. Δεν ξέρω αν το βλέπετε εσείς, έχω αυτή την άποψη, να βάλουμε τρεις πτυχές προς συζήτηση, σημαντικές. Τη διεύρυνση εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης της παλιάς οδηγίας για την κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων. Πρώτο αυτό. Δεύτερο, κυρώσεις, πολιτική κυρώσεων όταν δεν υπάρχει σεβασμός των δικαιωμάτων στις χώρες ε, προς τις επιχειρήσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτον να δοθούν και φορολογικά κίνητρα και να προωθηθούν οι βέλτιστες πρακτικές που έχουν εφαρμοστεί. Νομίζω ότι ίσως μπορούμε να συζητήσουμε αυτά τα θέματα. Ίσως μπορούμε να εντοπίσουμε έναν κοινό δρόμο που μπορούμε να ακολουθήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Παντσέρη, κύριε Παγαθόρτον Τούα. Ευχαριστώ τηλεγραφικά για να μην στερήσω χρόνο από άλλους συναδέλφους ή άλλους ε, που θέλουν το λόγο. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω το Προεδρείο και την Πρόεδρο που προκάλεσε αυτή τη συζήτηση και οργάνωσε αυτή τόσο σημαντική ενδιαφέρουσα ακρόαση. Και πράγματι, ε, παρότι ήταν πολύ δύσκολο, καταφέρατε να οργανώσετε αυτή την εκδήλωση, γι' αυτό και σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Έχουμε παγκοσμιοποιημένο οικονομικό κόσμο. Θα πρέπει λοιπόν να αναζητήσουμε ε, κοινούς τρόπους για την ε, ε, πράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Είναι κάτι που πρέπει να γίνει. Δεν είναι θέμα μόνο δικαιοσύνης. Πρέπει να βρούμε αποτελεσματικούς τρόπους πράσπισης αυτών των δικαιωμάτων και πρέπει να το κάνουμε και αν θέλετε καθαρά εγωιστικά όχι μόνο να ξεκινάμε συζητήσεις και διάλογο, αλλά να βρούμε ε, και αποτελεσματικές μεθόδους αφού εντοπίσαμε την αναγκαιότητα αυτή. Είμαι μέλος ε, καινούριο ε, της, του Κοινοβουλίου, είμαι στην Επιτροπή αυτή και στην Επιτροπή ΔΕΒΕ και πρέπει νομίζω να εκμεταλλευόμαστε τις πληροφορίες και όπως αυτές που μας δώσατε σήμερα για να μελετήσουμε και να δούμε τα, στα επόμενα σχέδια δράση και προγράμματα εργασία, πώς θα εντάξουμε την ανάγκη αυτή και πώς θα ζητήσουμε και από τις ε, διάφορες πολιτικές να ασχοληθούν και με τους άλλους απόλυτα θεμητούς στόχους, αλλά και με αυτούς για την πράσπιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν, τα πάρα πολύ πολύτιμες οι πληροφορίες αυτές και θα προσπαθήσουμε με αποτελεσματικό τρόπο και εμείς να τις, ε, να εντάξουμε ε, στις πολιτικές μας εγκάρσια. Και στην Επιτροπή Ανάπτυξης όμως, κοινωνική εταιρική ευθύνη, θα επαγρυπνούμε και όλη αυτή τη ροή πληροφοριών και τους στόχους θα τις εντάξουμε όλα αυτά, θα εντάξουμε όλα αυτά στο δικό μας ε, πρόγραμμα εργασίας. Σας ευχαριστώ κύριε Παγαθαρτοντώ. Σίγουρα ένας από τους στόχους, λέει πρόεδρος, με αυτή την ακρόαση και με την όλη δουλειά που επιτελούμε είναι να δώσουμε αυτό το μήνυμα, αυτή την πρωτοβουλία, να την μεταλαμπαδεύσουμε και σε άλλες ε, επιτροπές, γιατί πράγματι πρέπει να είναι οριζόντια η προσπάθεια. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές Μας έδωσαν πολύ ενδιαφέροντα μηνύματα. Έχω κάποια ερωτήματα. Πρώτα απ' όλα, για τις οργανώσεις που εκπροσωπούν οργανώσεις των δικαιωμάτων σε διάφορα επίπεδα. για να Η αναπτυξιακή πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε ποιο βαθμό παρέχει ορατή, τόσο σημαντική ενίσχυση επιτόπου. Μιλάμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις εργασίας, θέλουμε να επιτύχουμε την ευαισθητοποίηση της κοινή γνώμης. Πρώτο αυτό. Δεύτερον, για τους ε, εκπροσώπους ε, των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Αν κατάλαβα καλά, είπατε ότι κατά κάποιο τρόπο οι Ηνωμένε Πολιτείε ε, οι επιχειρήσει τους έχουν καλύτερα αποτελέσματα, έχουν μια πιο έτσι, καλή γραμμή υιοθετή που μπορεί να ακολουθηθεί. Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, οι ενό επιχειρήσεων, έχουν επαφές με τους Αμερικανούς ομολόγους ε, και πώς μπορούν να, να υποφεληθούν από τις βέλτιστες πρακτικές ή τις συμβουλές που μπορούν να λάβουν από αυτούς. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, θα δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Μαριό Βερονίκ. Το επιθετό σας είναι αυτό. Α, όχι, το δεύτερο όνομα σας. Μάλιστα, στην κυρία Μαριό Βερονίκ Καντιέ, λοιπόν. Θα σας δώσω σας το λόγο και έπειτα θα μιλήσουν οι εκπρόσωποι της Κομισιόν και της ΕΙΕΔ. Ε, ευχαριστώ πολύ. Σε σχέση με, τα, με τις διαθέσιμες κατευθύνες γραμμές και το πλαίσιο, θα συμπληρώσω φαντασμό Ρώμα, αλλά ε, έχουμε τις, ευρωπαϊ... έχουμε τις ευρωπαϊκές κατευθυντήριες ε, γραμμές. Στα ανθρώπινα δικαιώματα υπάρχει ανακαίωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπή Υποαναθεώρηση. Πρόκειται να επεκδοθούν κατευθυντήριε γραμμέ για τα εθνικά προγράμματα δράση, για την υλοποίηση των κατευθυντήριων αρχών των ΗΠΑ και άρα βλέπετε ότι υπάρχουν μηχανισμοί διαθέσιμοι. Πρέπει απλώ να υπογραμμίσουμε το γεγονό ότι χρειάζεται να υπάρξουν κατευθυντήριε γραμμέ, διότι όπω βλέπετε η υλοποίηση των κριτηρίων αρχών των Ηνωμένων Εθνών σε διάφορες χώρες και τις Ηνωμένες Πολιτείες παρουσιάζει κενά. Κάτι γίνεται, αλλά ακόμα υπάρχουν σημαντικά κενά, κενά που πρέπει να συμπληρωθούν και είναι σημαντικό να δερματίσει το ρόλο της η Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να προσφέρει κατευθύνσεις και καθοδήγηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα το Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Αν έχετε κάτι να προσθέσετε κι εσείς. Ναι, για το θέμα αυτό της καθοδήγησης. Εξασφαλίστηκε νομίζω αρκετή σαφήνεια για τις επιχειρήσεις UNGPs, οι κατευθύνες δηλαδή αρχές των ε, Ηνωμένων Εθνών οι τομεακές επίσης ε, κατευθυντήριες γραμμές που έχει επεξεργαστεί η Επιτροπή Υπάρχουν όλα αυτά. Ίσως θα μπορούσατε να μας κατηγορήσετε πριν από λίγο καιρό ότι είναι ήταν πρόημο να νομοθετήσουμε γιατί δεν ήταν σαφή ακόμη η κατάσταση α, και οι προσδοκίες. Αλλά νομίζω ότι τώρα πια μπορούμε να έχουμε ένα οδηγό τις κρατητήρης γραμμές των Ηνωμένων Εθνών. και πια ξέρουμε τι χρειάζεται να κάνουμε επιχειρήσεις και μπορούμε να πάρουμε μια πιο αποφασιστική δράση και να περάσουμε στην υλοποίηση, την πρακτική. Νομίζω ότι πλέον ε, οι κατευθυντήριες γραμμές σε θελοντικά αυστηρά βάση αποδεικνύουν ότι είναι περιορισμένες ε, περιορισμένος ο αντικτυπός τους και άρα θα πρέπει να περάσουμε σε μια ρυθμιστική επιλογή. Επίσης ε, για τον κύριο Παντσέρη που αναφέρθηκε στο σεβασμό των ανθρωπινών δικαιωμάτων. Νομίζω ότι θα πρέπει να μιλήσουμε και για το μη σεβασμό των ανθρωπινών δικαιωμάτων για τις επιχειρήσεις. Έχει ένα κόστος αυτό λοιπόν ως προς την δημόσια του εικόνα, ως προς τους πόρους, ως προς, την, ε, προς νομικά ζητήματα, ως προς τις δραστηριότητες τους ορισμένες περιοχές, οι οποίες ε, δυσχεραίνουν λόγω συγκρούσεων με τις τοπικές κοινωνίες ή διότι προκύπτουν προβλήματα όπως αυτό, τραγωδίες όπως αυτή της Ράνα Δηλαδή έχει κόστος και για την επιχείρηση αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε τους εκπροσώπους από την Επιτροπή Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων και η κυρία που είναι υπεύθυνη για την κοινωνική ευθύνη. Η κυρία Σοφή Μίλλερ, παρακαλώ, πέντε λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλους. Και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που είχατε την πρωτοβουλία αυτή τη ακρόαση και θέσατε το θέμα τη εταιρική ευθύνη και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη μερίσια σα διάταξη, θα ήθελα να σα δώσω μια πολύ σύντομη επισκόπηση του, των θέσεων τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και του προγράμματό τη για την κοινωνική ευθύνη. Είδαμε σήμερα από τη συζήτηση ότι είναι ένα θέμα πολύ περίπλοκο, είναι ένα θέμα το οποίο απαιτεί και την ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων και πολύ τομεακή συνεργασία και γι' αυτό θα μου επιτρέψετε να δώσω το λόγο και στον συνάδελφο από την Υπηρεσία εξωτερική Δράσεω και από την Γενική Διεύθυνση Απασχόληση για να σα δείξουμε και την εξωτερική διάσταση των, ε, ειδικά για τα δικαιώματα των εργαζομένων. Ποια είναι λοιπόν η πολιτική της Επιτροπής για την εταιρική ευθύνη, σε τι αποσκοπεί, ε, αποσκοπεί στην ανάπτυξη σημαντικών και σοβαρών ε, δράσεων σε επίπεδο κρατών μελών. Έχουμε νομίζω ήδη αρκετά ε, σαφή νομοθεσία πολλές φορές άκαμπτη νομοθεσία στα θέματα αυτά θα σας εξηγήσω εν τι πορεία και τι συγκεκριμένα σημαίνει αυτό ε, για δε τις στρατηγικές που αναφέραμε από το 2012, όταν μιλάμε για εταιρική ευθύνη, θέλουμε οι εταιρείε να αναλαμβάνουν τις ευθύνες για, την, ε, για τον αντίκτυπο των δράσεών τους στην κοινωνία. Αυτό είναι περίπλοκο. Μιλάμε σήμερα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θέλουμε όμως και για το περιβάλλον να αναλάβουν την ευθύνη για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Για κάθε κοινωνικό θέμα, δεοντολογικό ή δικαιώματα καταναλωτών. Λίγο πολύ αυτή είναι η γενική περιγραφή των καθηκόντων μας και θέλω να πω ότι η πολιτική μας δεν κοιτάει ούτε ένα συγκεκριμένο θέμα, ούτε ένα συγκεκριμένο τομέα. Αναφέρεται σε 21 εκατομμύρια ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και αφορά 21 εκατομμύρια ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Αυτό ίσως μπορούμε να το δούμε σαν μια προσπάθεια συμπληρωματική σε σχέση με τις επιμέρους πρωτοβουλίες που έχουν ξεκινήσει. Η γενική μας προσέγγιση λοιπόν είναι ότι θέλουμε οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να ενσωματωθούν στα διεθνή ε, πλαίσια. Μιλήσαμε για την τριμερή της Διεθνούς Οργανίσεως Εργασίας, για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην ΕΕ, για τον ΩΣΑ και τις ε, κατευθυντήριες γραμμές για τις επιχειρήσεις, για την ISO 26000, για το Global Compact. Όλα αυτά λοιπόν σε διεθνές επίπεδο συναποτελούν ένα πολύ στεναρό πλαίσιο το οποίο μπορεί να οδηγήσει επιχειρήσεις σε πιο υπεύθυνη δραστηριοποίηση. Έγινε λόγος και για συμπληρωματικές και εθελοντικές ρυθμίσεις. Συμφωνώ ότι είναι κέρια η σημασία ενός εφιού μείγματος Smart Mix. Έχουμε παραδείγματι από πλευρά της Επιτροπής για να αναφερθώ στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το 99% των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, των συνόλων των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Μια επιχείρηση λοιπόν η οποία απασχολεί πέντε εργαζομένων ίσως να μην την έχει απασχολήσει το ζήτημα των ανθρώπινων δικαιωμάτων ε, αν απασχολεί εργαζόμενους. Όμως θέλουμε και για τις μικρές και μεσές επιχειρήσεις να δώσουμε λύσεις ε, σημαντικές, ε, εφόσον αυτές είτε προμηθεύονται, είτε δρούν, είτε έχουν κάποια άλλη δραστηριότητα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης για το ρυθμιστικό ζήτημα και αναφέρθηκε, αναφέρθηκε το παράδειγμα των ΗΠΑ που έχουν κατά πάσα πιθανότητα ηγετική θέση σε σχέση με την Μιανμάρ, αλλά έχουμε εμείς μια υποχρέωση για την λογοδοσία για τις δραστηριότητες σε όλες τις χώρες ανά τον κόσμο. Αναφέρεται στις μεγάλες επιχειρήσεις, γιατί έχουμε τον περιορισμό από το Συμβούλιο, αλλά δεν πιστεύουμε ότι αποτελεί την ορθή προσέγγιση το να επιβάλλονται περιορισμοί μόνο για μία χώρα χώρα. Ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι και τα εργασιακά δικαιώματα είναι οικουμενικά και εξίσου οικουμενική πρέπει να είναι και η προσέγγιση μας. Αυτό θέλουμε να το δούμε, να το αντιληφθούν και οι επιχειρήσεις, γιατί υπάρχουν οι οδηγίες εκείνες για τη λογοδοσία, στις οποίες εφαρμόζονται αυτές οι αρχές. Και επίσης θέλουμε και τις οδηγίες τις σχετικές με τις προμήθειες να ενσωματωθούν αυτές οι αρχές υιοθετήθηκαν από το Κοινοβούλιο τον Ιανουάριο και μπορούν οι δημόσιες αρχές να απορρίψουν προμήθεια, σύμβαση προμήθειας ή και να την αναστείλουν, να αναστείλουν τη λειτουργία της εφόσον υπάρχουν ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αυτό βέβαια αφορά και την δραστηριοποίηση εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναφερθήκαμε επίσης στην αναπτυξιακή βοήθεια. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, παραδείγματι, έχει καταστήσει, έχει διατυπώσει σαφείς προϋποθέσεις ανθρωπινών δικαιωμάτων και τις έχει καταστήσει οι υποχρεωτικές δεσμευτικές δηλαδή για τι δραστηριότητε των επιχειρήσεων που χρηματοδοτεί εκτός Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει δηλαδή πρόοδο. Επίσης θα έχω, μπορούσα να πω ότι έχουμε ένα νομικό πλαίσιο που επιτρέπει οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις με τον κανονισμό Βρυξέλλες 1 να επιτρέπει να προσαχθούν ενώπιον Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου εφόσον δεν τηρούν του κανόνε που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πολύ συγκεκριμένε προποθέσει. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει διατυπώσει σαφέστατα του όρου αυτού, αλλά πάντω μπορεί μια τέτοια διαδικασία να οδηγήσει σε προσαγωγή μιας επιχείρησης ενώπιον ενός ευρωπαϊκού δικαστηρίου. Αυτά λοιπόν ε, εν γέννη. Υπάρχουν αρκετά πράγματα που μπορούμε να συζητήσουμε φαντάζομαι. Έχουμε, την ευθύνη της, ε, έχουμε το θέμα της λογοδοσίας για την κοινωνική ευθύνη. Η διεθνής αλυσίδα προμηθειών είναι ένα ζήτημα που πρέπει να προχωρήσει ιδιαίτερος. Και βέβαια και οι συζητήσεις θα διδραματίσουν πολύ σημαντικό ρόλο. Ευχαριστώ. Και τώρα ο κ. Ρικάρδο Σέρι, επικεφαλής της, ε, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης που έχει το λόγο για πέντε λεπτά. Ευχαριστώ. Και εγώ, όπως και συνάδελφος, θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου για τη συζήτηση. Ποικιλόμορφη, πολλές φωνές, πολλές απόψεις, ζητήματα τίθενται και εν γέννη εμπίπτουν στο ευρύτερο πλαίσιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τέθηκαν ζητήματα. Αναφέρθηκαν συγκεκριμένες χώρες. Βιρμανία, Καμπότζη, παραδείγματο χάρη, Μπαγκλαντές και άλλες. Θα ήθελα εν συντομία να εξηγήσω τι προσπαθούμε να κάνουμε όσον αφορά την υπηρεσία εξωτερικής δράσης και δράτω με τις ευκαιρίες να εστιαστώ στις κατευθυντήριες γραμμές. Απαντώντας έτσι σε ερωτήσεις της κυρίας Λόχμπιλερ. Αλλά και άλλα θέματα που τέθησαν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση από την αρχή ήταν ένθερμη υποστηρίκτρια των κατευθυντήριων γραμμών. Αυτές οι γραμμές είναι προϊόν γενικής συνενέσεως. Σε επίπεδο κυβερνητικό, με συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα και της κοινωνίας των πολιτών. Εκπληκτικό επιτεύγμα θα έλεγα. Δεν ήμουν εκεί στη συζήτηση, αλλά οι συνομιλίες για δεσμευτικό μέσο κράτησε δεκαετίες. Θέλαμε να θεσπιστούν πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πολλέ προσπάθειε είχαν γίνει κατά το παρελθόν και απέτυχαν. Οι κατευθυντήριε γραμμέ είναι έξοχο επίτευγμα. Του 2011, Προτριετία. Αυτό λέγαμε πάντα, ότι είναι καλό επίτευγμα που χρήζει επεξεργασίας. Αυτό κάναμε μέχρι τώρα. Το ακούσατε σήμερα και θα το ακούσετε και στο μέλλον. Περιπλοκότατο ζήτημα. Άρα πρέπει να καταλάβουμε οι ίδιοι τι πρέπει να κάνουμε και που υπάρχουν κενά. Όπως αναφέρθηκε, υπάρχει ένα έγγραφο που συντάσσεται, έγγραφο πολιτικής που αναλύει την κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα μελλοντικά βήματα σημαντικό για μας. Και χρειάζεται μια ενδελεχή ανάλυση για να προχωρήσουμε. Με συνέπεια είχαμε μια ομόφωνη θέση στη Γενέβη, στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Δηλαδή, θέλουμε να ξεπεράσουμε τα παρόντα πλαίσια των κατευθυντηρίων γραμμών. Να προχωρήσουμε για συνθήκη τώρα σε αυτή τη φάση ίσως να είναι κάτι αντιπαραγωγικό. Εκεί βασίστηκε η θέση μας, που εξηγήθηκε δημοσία. Υπήρχε ξανά διχασμός στο Συμβούλιο. Μια διακυβερνητική ομάδα θα επεξεργαστεί το θέμα της συνθήκης, θα συνεδριάσει τον Ιούνιο στη Γενέβη θα παρακολουθήσουμε εκ του σύνεγγες τις εξελίξεις, θα θέλαμε να γνωρίζουμε την πορεία που θα ακολουθηθεί. Αυτό που θέλουμε τώρα είναι να επεξεργαστούμε την εφαρμογή των κατευθυντηρίων γραμμών των Ηνωμένων Εν συντομία, συνοψίζω τα όσα κάνουμε. Συζητούμε τα θέματα αυτά στα πλαίσια του διαλόγου μας περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων πολλές χώρες. Πρόσφατα έγινε συζητήσει με Βραζιλία και Μεξικό. Έχουμε τον κύριο Λαμπρινίδη, τον ειδικό μας εκπρόσωπο, που καταβάλει άοκνες προσπάθειες στις συζητήσεις με τους εταίρους. Προωθούμε σεμινάρια σε συνεργασία με τίτες χώρες. Πιστεύουμε σε περιφερειακές ομάδες και συμμετοχή των περιφερειακών φορέων Μόλις πριν μια εβδομάδα συναντηθήκαμε με την Αφρικανική Ένωση στην Αντίσα Μπέμπα. Διοργανώσαμε σεμινάριο όσον αφορά τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΗΕ. Τους είπαμε τι κάνουμε στον ΟΗΕ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση διορθώνει ο μιλητής. Κυρίως προετοιμάζοντας τα εθνικά σχέδια δράσης των κρατών μελών και συμφωνήσαμε με την Αφρικανική Ένωση να συνεχιστεί η προσπάθεια. Ε, θέλει ο φορέας αυτός να συμμετάσχει ενεργά στην επεξεργασία των κατευθυντήριων γραμμών και μαζί με τον ΟΗΕ που συμμετείχε στο σεμινάριο της Αντίσα Μπέμπα θα συνεχιστεί συνεργασία για να καταλήξουμε σε κάποια χρηματοδότηση της Αφρικανικής Ενώσεως για να εφαρμόσουν τις κατευθυντήριες γραμμές στο σύστημά τους και για να υποστηρίξουμε τα κράτη-μέλη της Αφρικανικής Ένωσης να κάνουν κάτι παρόμοιο και να ετοιμάσουν εθνικά σχέδια δράσης. Είναι ένα παράδειγμα αυτό του τι μπορούμε να κάνουμε και τι θα εξακολουθούμε να κάνουμε την επόμενη τριετία τουλάχιστον σε συνεργασία με περιφερειακούς φορείς και τους εταίρους μας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε εμείς, κύριε Σέρη. Φυσικά και εμείς θα σας παροτρύνουμε να συνεχίσετε σε αυτή την πορεία και εμείς θα εξακολουθήσουμε να αποδίδουμε τη μέγιστη προσοχή στο έργο και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των Γενικών της Διευθύνσεων και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Θα δώσω τώρα στον κύριο Ρούντι Ντελαρή το λόγο που είναι ο επικεφαλής μονάδας για τις εξωτερικές σχέσεις της ΓΔ Πασχόλης Κοινωνικές Υποθέσεις. Έχετε και εσείς πέντε λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε, θέλω και εγώ να σας συγχαρώ όπως προλαλήσατε συναδελφοί μου για την εκλογή σας και τα μέλη της Επιτροπής σας. Να ευχαριστήσω επίσης και τους ομιλητές για τις πληρέστατες παρουσιάσεις τους. Όπως είπαν οι συνάδελφοί μου, θα ακολουθήσουμε μία διεπιστημονική προσέγγιση. Θέλουμε να προωθήσουμε τα δικαιώματα των εργαζομένων και ε, να τα εντάξουμε στις ε, διάφορες πολιτικές μας και με συγκεκριμένες ενέργειες και με συνεργασία με τα άλλα θεσμικά όργανα και με τα κράτη-μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους σε όλα τα επίπεδα, επιχειρήσεις και των πολιτών. Και στο πλαίσιο διεθνών οργανισμών όπως η Διεθνή Οργάνωση Εργασίας, ο όσα και στο πίσω αλλά και σε συνεργασία με αυτού, του οργανισμού. εργαζόμαστε. Αυτή λοιπόν η συνολική προσέγγιση έρχεται ε, να συνδεθεί ε, στο στόχο αυτό για την ε, στήριξη των ανθρώπινων δικαιωμάτων και δικαιωμάτων εργαζομένων στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης. Είναι προσπάθειες που είναι σε εξέλιξη, το Κοινοβούλιο έχει στηρίξει τις προσπάθειες, πρέπει να κάνουμε ακόμη πολλά ακόμα. Συγκεκριμένα παραδείγματα και του τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τα εργασιακά πρότυπα, τα δικαιώματα των εργαζομένων, θα τα βρείτε σε μια ανακοίνωση του Φεβρουαρίου του 2014 από τη ΓΔ Απασχόληση. Αν δεν έχουν διατεθεί, θα σα διατεθούν ήδη ορισμένα αντίτυπα αυτή τη ανακοίνωση. Θα ήθελα να σα δώσω κάποια συγκεκριμένα παραδείγματα για να σα δείξω πώ λειτουργούμε. Η διεθνή ε, συνεδρίαση εργασία ε, του ΔΟΕ έβγαλε ένα πρωτόκολλο για την καταναγκαστική εργασία Πολύ σημαντική πρωτοβουλία, υπήρξε πολύ καλός συντονισμός και από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγκρίναμε και στηρίξαμε αυτή τη, αυτό το πρωτόκολλο και επίσης ε, πρόσφατα παρουσιάσαμε πρόταση στο Συμβούλιο ζητώντας από τα κρατη να ε, εγκρίνουν αυτή την πρόταση και ζητώντας να εγκριθεί αυτή, αυτό το πρωτόκολλο στο δυνατό. Η πρόταση ήδη ε, υποβλήθηκε το Σεπτέμβριο συγκεκριμένα Γρήγορα δράσαμε και γιατί, γιατί θέλαμε τα κράτη-μέλη να δώσουν το καλό παράδειγμα και για τον υπόλοιπο κόσμο, θέτοντας σε εφαρμογή αυτό το πρωτόκολλο. Το Κοινοβούλιο βέβαια τώρα και το Συμβούλιο πρέπει να εγκρίνουν αυτή την πρόταση και ελπίζουμε αυτό να γίνει σύντομα. Η απαγόρευση της καταναγκαστικής εργασίας βέβαια είναι ε, μία ε, βασική ε, αρχή, είναι ένα από τα βασικά θεμελιώδη δικαιώματα της χάρτης του ΟΗΕ για τα, για τα δικαιώματα εργασίας. Έχουν οκτώ πρότυπα, έχουμε οκτώ τέτοια πρότυπα από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας, τα έχουν προσχωράψει και δεχθεί όλα τα κράτη-μέλη. Και αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να συμπεριλάβουμε τις ρήτρε αυτές ε, στις ε, συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών. Έχουμε το κεφάλαιο αυτό που περιλαμβάνουμε τις, ε, τα εργασιακά αυτά πρότυπα και κανόνες και δεσμεύσει και από τις δύο πλευρές. Πέραν των δεσμεύσεων όμως, σε αυτές τις συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών μιλάμε για την αξιοπρεπή εργασία για όλους, για την επικύρωση, πρόθεση της επικύρωσης άλλων επικαιροποιημένων συμβάσεων του, της ΔΟΕ, για την επιθεώρηση εργασία, κοινωνική ασφάλεια κτλ. κτλ. Επομένως, α, να πω και κάτι ακόμη. Πέραν αυτών των ε, συμφωνιών ε, υπάρχει ένα σύστημα παρακολούθηση. Συμμετέχει η κοινωνία των πολιτών και η κοινωνική Εταιρεία σε αυτή τη διαδικασία. Είναι μια νέα γενιά συμφωνιών βέβαια και για μα είναι καινούργιο αυτό. Γι' αυτό και παρακολουθούμε από κοντά τα πράγματα. Υπάρχει και το γενικευμένο σύστημα προτιμήσεων που είναι ένα εμπορικό μηχανισμό. Έχουμε και το γενικευμένο σύστημα ΣΥΝ, το οποίο ε, έχει ω προαπαιτούμενο την έγκριση αυτών των οκτώ εργασιακών προτύπων και άλλων συμβάσεων τη ΔΟΕ και είναι προαπαιτούμενο, παραλαμβάνω, για προσχώρηση σε αυτό το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων ΣΥΝ. Υπάρχει το εποπτικό σύστημα της ΔΟΕ, Υπάρχουν πορίσματα και από άλλου διεθνεί οργανισμού. και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ιδιαίτερα δραστήρια στο πλαίσιο του διαλόγου. Παραδείγματος χάρη υποπτική ε, βοήθεια. Είναι σημαντικέ υποθέσει που μα έχουν απασχολήσει για τα δικαιώματα των εργαζομένων, όπω το παρελθόν τη Μιανμάρ, ε, Λευκορωσία, Ουσμπεκιστάν και άλλε χώρε. Η Συμφωνία ελευθερου εμπορίου περιλαμβάνουν και άρθρα συνεργασίας για θέματα απασχόλησης ε, κοινωνικής πολιτικής. Εκεί εντάσσονται και τα δικαιώματα των εργαζομένων. Πρέπει να εφαρμόζονται στην πράξη. Τώρα περνώ σε δύο καινοτόμες προσεγγίσεις. Το σύμφωνο βιωσιμότητας του Μπαγκλαντές είναι ένα παράδειγμα. Θέλω να τονίσω ότι πρόκειται για μια καινοτόμο προσέγγιση γιατί. Διότι πρόκειται για εταιρική σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης του Μπαγκλαντές ως τρίτης χώρας, της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας αλλά και των Ηνωμένων Πολιτειών που έχουν προσχωρήσει σε αυτό το σύμφωνο. Επίσης θέλω να σας πω ότι αποτέλεσμα ε, αυτή τη διαδικασία ήταν πολλές βελτιώσεις ε, ε, στα δικαιώματα των εργαζομένων και στι συνθήκε υγιεινή και ασφάλεια στον χώρο εργασία των Μπαγκλαντέ. Θα γίνουν πολλά ακόμη. Έχουμε μία συνεδρία στον Οκτώβριο στι Βρυξέλλε. Αυτή η καινοτόμω προσέγγιση θα μπορούσε να βρει μιμητέ και σε άλλες περιπτώσεις, να εξαχθεί, να αναπαραχθεί. Υπάρχει και η συμφωνία, το ακόρτ, ε, όπως λέμε, το επέγραψαν επιχειρήσεις ε, και τα συνδικάτα και έχουμε και την πρωτοβουλία για την ε, αποζημίωση των θυμάτων. Για το ακόρτ, αυτή τη συμφωνία πρέπει να σας πω ότι ήταν ηγετική στάση που επέδειξαν ε, οι ευρωπαϊκέ επιχειρήσει, πολύ περισσότερο από ό,τι από επιχειρήσει άλλων χωρών. Μια άλλη καινοτόμα προσέγγιση. Η πρόεδρο διακόπτει τον ομιλητή. Ναι, ναι, να ολοκληρώσω, να ολοκληρώσω. Θαλάσσια σύμβαση και αυτή καινοτόμα προσέγγιση είναι, πιστεύω, διότι συνδυάζει τα ευρωπαϊκά με τα διεθνή συστήματα επιβολής Τη νομοθεσία και έτσι αντισταθμίζει κάποια κενά που είχαμε με πλοία που κυκλοφόρησαν με σημαία ευκαιρία. Ε, στους διάλογους μας με τρίτες χώρε για θέματα απασχόληση κοινωνικών υποθέσεων όπω Κίνα, Ινδία, μιλούμε για την υγειακή ασφάλεια στην εργασία, μιλούμε για τα θέματα κοινωνική προστασία και βέβαια και στην πολιτική γειτονία ε, αναφέρομαι αυτά τα ζητήματα και για την επικύρωση και την ε, εφαρμογή των βασικών στρατηγικών ε, και προτύπων εργασιακών ε, του, της ΔΟΕ. Αυτά είναι προτεραιότητά μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, συνεισφέρει λοιπόν και αν δείτε και τα απορίσματα τα τελευταία του Συμβουλίου Υπουργών θα δείτε ότι είναι ένα σημαντικό θέμα για μας. Και φυσικά θα συνεχίσουμε το διάλογο και τη συνεργασία μας με εσά. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ πολύ. Δεν είναι η τελευταία φορά, δεν είναι η τελευταία φορά που έχουμε αυτή τη συζήτηση, αυτό το διάλογο για το θέμα αυτό. Είναι η πρώτη φορά, είναι η απαρχή μια σειρά από ε, τέτοιε ευκαιρίε που θα μα δοθούν και στη συνέχεια. Ήταν όμω πολύ χρήσιμη αυτή η ακρόαση για όλους μας. Ε, θα συναντηθούμε πάρα πολύ σύντομα με όλους. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους και ε, όλες όσες ήρθατε εδώ για να μας ε, παρουσιάσετε τη δική σας εμπειρία από την επιτόπου δουλειά που κάνετε. Ήταν πάρα πολύ σημαντική συνεισφορά και για τους βουλευτές που είμαστε εδώ, αλλά και για τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Μόλις ξεκινάμε τον αγώνα μας, τη μάχη μας, και ελπίζω να μπορώ να βασιστώ σε όλους σας για τους επόμενους μήνες. Ευχαριστώ πολύ όλες και όλους και εδώ λίγη ακρόαση. Όσοι, μπορώ, έχετε την ε, άδεια να είστε παρόντες, ε, εξοδοτήστε να είστε παρόντες στη συνεδρία του Ευρωπαϊκού Προεδρείου, να σας πω ότι αρχίζουμε στις 11.30.